Okay, colleagues, we are going to make a start. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε αργήσει ήδη κάποια λεπτά να φροντίσουμε ο χρόνος που καθυστερήσαμε να αφαιρεθεί από το δικό μου χρόνο ομιλίας. Ε, χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ σήμερα και ε, προεδρεύω αυτή τη ε, ακρόαση. Θα ήθελα ιδιαίτερως να καλωσορίσω από πλευρά της Επιτροπής μας τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος έχει διοριστεί για Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων. Κάποιοι από εσά ήσασταν εδώ χθε το βράδυ. Για όσου ε, δεν είσαστε εδώ πέρα, θα ήθελα να εξηγήσω εκ νέου τη διαδικασία. Το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον ε, άρθρο 118 και παράρτημα 16 του κανονισμού, προετοιμάζει τι ε, ακροάσει αξιολογώντας όλους τους υποψηφίους ε, επιτρόπους βάσει της γενικών τους ικανοτήτων, τη δέσμευσή τους σε ευρωπαϊκά ζητήματα και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Επίσης, το Κοινοβούλιο αξιολογεί την κατανόηση του χαρτοφυλακίου του υποψηφίου και τις ε, επικοινωνικές του ικανότητες. Και αυτό το σκοπό λοιπόν εξυπηρετεί η σημερινή ακρόαση, να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Να σας ενημερώσω ότι η ακρόαση αυτή μεταδίδεται ε, ζωντανά στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Europe by Satellite. ορίζουμε λοιπόν και όσους μας παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου ή μέσω του Europe by Satellite, μέσω δορυφόρου. Ε, οι μαγνητοσκοπήσεις επίσης θα διατεθούν μετά την ακρόαση από όσους το ζητήσουν. Για την για σημερινή ακρόαση έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες. Ε, όλοι έχουν χρονική πίεση, αλλά σας παρακαλώ να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα για να μπορούν να σας παρακολουθούν και οι διερμηνείς. Είναι μάλιστα σήμερα και η Διεθνή ημέρα της μετάφρασης. Άρα ευχόμαστε σε όλους τους διερμηνείς μας ε, καλή ημέρα της μετάφρασης και χαιρόμαστε πολύ που τους έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα και από εμάς. Έχουμε αποστείλει κάποιες γραπτές ερωτήσεις στους υποψηφίους, στον υποψηφίο επίτροπο και έχει απαντήσει. Έχετε αντίτυπα των απαντήσεων και διατίθενται άλλωστε και στην αίθουσα για, του, για τους βουλευτές. Να σας εξηγήσω τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Θα ξεκινήσει ο κ. Στυλιανίδης με μία δήλωση 15 λεπτών κατά ανώτατο όριο. Και το βασικό τμήμα της ακρόασης θα αποτελείται, όπως και χθε το βράδυ, από 45 ερωτήσεις. Στον πρώτο γύρο κάθε πολιτική ομάδα θα έχει μία ερώτηση ενός λεπτού και ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει 1,5 λεπτό για να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Μετά την απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου. Θα υπάρχει ενδεχομένω ε, ε, δεύτερη ερώτηση, υπερέτηση για 30 λεπτών και απάντηση ενό λεπτού. Τέσσερα λεπτά λοιπόν σύνολο για τον πρώτο γύρο. Όλε οι υπόλοιπε ερωτήσει θα διαρκέσουν ε, τρία λεπτά σύνολο. Μία, ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Συνάδελφοι, παρακαλώ να έχετε υπόψη τα χρονικά περιθώρια, το χρονικό πλαίσιο, γιατί δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τον προβλεπόμενο χρόνο. Επίσης θα έχουμε ερωτήσεις από τις δύο επιτροπές που έχουν προσκληθεί στην ακρόαση γιατί εμπίπτουν ε, στον τομέα των αρμοδιτήτων τους ε, το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου επιτρόπου είναι η Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και μετά θα ανοίξει η συζήτηση για ερωτήσεις από τις πολιτικές ομάδες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα. Κυρία Στυλιανίδη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά μάξιμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματική τιμή η παρουσία μου εδώ σήμερα ως υποψήφιος επίτροπος στην ανθρωπιστική βοήθεια και την διαχείριση των κρίσεων. Είναι μεγάλη τιμή που προτάθηκα για αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι στην καρδιά των πανανθρωπίνων αξιών έχω πλήρη συνέστηση της τεράστιας ευθύνης. Είμαι ενώπιόν σας ως συνάδελφος, ως πολιτικός που απευθύνεται σε πολιτικούς. Δουλειά μας είναι να λαμβάνουμε αποφάσεις. Συχνά δύσκολες, πολύ δύσκολες αποφάσεις. Ένας πολιτικός είναι σε συνεχή πάλι με την ιστορία και είμαστε υπόλογοι προς τις επόμενες γενναίες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όραμα, πολιτικό θάρρος και αξιοπρέπεια. Ευθύνη μου είναι να παράσχω ε, την ε, ηγεσία που θα επιτρέψει το όραμα αυτό να γίνει αποτελέσματα επιτόπου. Οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια αυξάνονται καθημερινά. Συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή, καταστροφές θεμάτων υγείας, απόλυτη φτώχεια και πείνα είναι τα κύρια αίτια της αύξησης αυτών των αναγκών. Το, τα τρομερά γεγονότα καταδεικνύουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Μέχρι το τέλος του 2013, 51 εκατομμύρια άτομα ήταν εσωτερικοί εκτοπιστέντες λόγω συγκρούσεων και κατά μέσο όρο 32.000 άτομα εκτοπίζονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Πάνω από 8.000 παιδιά πεθαίνουν από υποσυτισμό και περίπου 3.000 πεθαίνουν τη μέρα που γεννώνται. Έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τώρα, όχι αργότερα. Σήμερα, όχι αύριο. Γνωρίζω τι σημαίνει να ζει κανείς κατάσταση σειράξεως. Να μην έχει καταφύγιο. Να μην έχει τα βασικότερα. Να λύσει φόβο. Να ζει σε φόβο, συγγνώμη. Και να του έχει αφαιρεθεί η αξιοπρέπειά του. Ως παιδί και κατόπιν ως έζησα τα δεινά του λαού της Κύπρου των Ελληνοκυπρίων και των Τούρκοκυπρίων. Έζησα το πόνο της εξορίας. Κατάλαβα στο πετσί μου τη σημασία και την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω να είμαι σαφής. Οι επιπτώσεις των σειράξεων δεν σέβονται εθνότητα ή θρησκεία. Φύγουν τους πάντες. Γέρους, νέους, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται σε ανάγκες, όχι πολιτικές σκοπιμότητες. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρομερές προκλήσεις στο εγγύς μέλλον. Πρώτα απ' όλα, θέλω να αποτίσω φοροτιμής ε, στους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και στην παροχή ανακούφισης. Κάθε μέρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλο, ανεξάρτητα από ταυτότητα, θρησκεία, εθνικότητα και ας φέρουμε στο μυαλό μας τη δολοφονία του Βρετανού εργαζόμενου στον ανθρωπιστικό τομέα David Haynes από το Ισλαμικό κράτος. Επίσης ας θυμηθούμε τη δολοφονία των, εκτά, των οκτώ θαραλέων ε, εργαζόμενων στον ανθρωπιστική, στην ανθρωπιστική βοήθεια και την υγεία που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τους κινδύνους του έμπολα. Αυτές είναι οι ε, οδυνηρές υπομνήσεις των κινδύνων που αντιμετωπίζουν αυτοί που εργάζονται για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά επίσης μας υπενθυμίζουν ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η παραβίαση των πιο βασικών θεμελιωδών αρχών που έχει καθορίσει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ο αριθμό των επιθέσεων κατά των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα έχει τετραπλασιαστεί από το 2003. Ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο ευαίσθητος λόγω της αυξανόμενης ε, συχνότητας και εντάσεως των θεομηνιών σε αναπτυγμένε χώρες, ακόμη και στην Ευρώπη. Συμβαίνουν επίση, για παράδειγμα, οι πλημμύρες που είδαμε στα Βαλκάνια τον περασμένο Μάιο ήταν οι χειρότερε για 100 χρόνια στην περιοχή. Η συλλογική ανταπόκριση της Ένωσης σε αυτήν τη θεομηνία ήταν άμεση και εντυπωσιακή. 23 κράτη-μέλη έδρασαν αλληλέγγυα υπό το συντονισμό του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης αποστέλλοντας εμπειρογνώμονες και ζωτική σημασία βοήθεια. Πέρα από τις ε, ανθρώπινες τραγωδίες, οι θεομηνίες έχουν επίσης επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την ε, αύξηση. Η διαχείριση των κρίσεων σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τον όλο κύκλο των θεομηνιών, περιλαμβάνοντας την πρόκληση και την ετοιμότητα. Την πρόληψη, συγγνώμη, και την ετοιμότητα. Και το κάνουμε αυτό στα κράτη-μέλη μα, βοηθώντα τα να μειώσουν του κινδύνους, αλλά και διεθνώ στα πλαίσια του πλαισίου χιόγκο για δράση. Η επικείμενη παγκόσμια διάσκεψη τον επόμενο Μάιο στο Σεντάι θα είναι μια ευκαιρία η πρόληψη και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των θεμενιών να είναι ισότιμες προτεραιότητες με την ανταπόκριση στις θεομηνίες. Οι απόψεις του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές και είμαι διατεθειμένος να συζητήσω μαζί σας εν ώψη αυτής της συνδιάσκεψης. Στον τομέα των σειράξεων η κατάσταση είναι δραματική. Για πρώτη φορά έχουμε τέσσερις κρίσεις επίπεδου τρία που είναι η υψηλότερη ταξινόμηση στο σύστημα των ΗΕ, Συρία, Ιράκ, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και Νότιο Σουδάν. Αλλά υπάρχουν και άλλες παρατεταμένες κρίσεις που εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Παλαιστίνη, Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό, Μαλή, Κολομβία, Μιανμάρ, για να αναφέρω μόνο κάποιες. Στη Συρία παρατηρούμε μία από τις μεγαλύτερες ε, ανθρωπιστικές καταστροφές που έχουν σημειωθεί ποτέ. Πολύ πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν θυγεί από τη σύραξη. 6,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα μισά είναι παιδιά, είναι εσωτερικά εκτοπιστέντες. Και ο αριθμός των προσφύγων έχει υπερβεί τα 3 εκατομμύρια. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα, όχι αύριο. Επιπλέον, έχουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα της επιδημίας έμπολα στη Δυτική Αφρική. Η έμπολα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τεράστιας κλίμακας θεομηνία. Είναι σαν να είναι ένας τυφώνας σε αργή κίνηση και επίσης είναι απειλή στην ε, πλανητική ασφάλεια όπως την καθορίζει το Συμβούλιο Ασφαλής των Εθνών πίσω από τις ε, ανισχυτικές στατιστικές για την τρομερή επέκταση του ιού βρίσκονται πραγματικές ανθρώπινες ζωές, λαοί και κοινότητες που θα χρειαστούν και ψυχολογική βοήθεια μετά την ανάκαμψη. Αυτές είναι πιεστικές κρίσεις, παρούσες και χρειάζονται αμέσως απάντηση, αλλά επίσης και μακροχρόνιο σχεδιασμό αυτή η μοναδική κατάσταση έχει θέσει το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα υποτρομερή πίεση. Είμαι πεπισμένος ότι η παγκόσμια ανθρωπιστική συνάντηση κορυφής το 2016 θα συμβάλλει στην βελτίωση των δυνατοτήτων του διεθνού συστήματος να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη βοήθεια, βοήθειας. Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση δυστυχώς δεν συμβάλλει στην ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για τη σταθερή και αποφασισμένη δέσμευση για την υποστήριξη ουσιαστικών επιχειρήσεων που σώζουν ζωές. Είναι επιτακτικό να αποφύγουμε διακοπές στις δραστηριότητες οικονομικής βοήθειας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε... Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία επαρκή ροή πληρωμών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Και τέλος, ορισμένα λόγια για το όραμά μου. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, αλλά εξίσου μεγάλη είναι η αποφασιστικότητα και ο ενθουσιασμός μου. Θέλω να ολοκληρώσω την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Καταρχήν, θα συνεχίσουμε με, το κύριο, με την κύρια εντολή μας έτσι ώστε να χορηγήσουμε βοήθεια στα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να φτάσει με πολύ λίγα και πολύ αργά. Ούτε μία φορά θέλω να συνεισφέρω έτσι ώστε οι υπεύθυνοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να μπορέσουν να παραμείνουν και να παραδώσουν ε, και δεν μιλώ μόνο για τις μεγάλες κρίσεις που βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά και για τις ξεχασμένες κρίσεις, όπως ονομάζονται. Δεύτερον, θα ήθελα να είμαι ο εκπρόσωπος των πλέον ευάλωτων, η φωνή εκείνων που δεν διαθέτουν φωνή. Θα εργαστώ την ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη, έτσι ώστε η φωνή εκείνων που πλήττονται να φτάσει στις τράπεζες λήψης αποφάσεων. Με θορύβησαν οι μαρτυρίες σε μία πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης για τη βία και την παρενόχληση των γυναικών της Συρίας που έχουν εκτοπιστεί. Οι γυναίκες και τα παιδιά βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και θα ήθελα να τους προσδώσω τη δέουσα προσοχή. Τρίτον, θα υπερασπιστώ τις ιδιαιτερότητες και τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει μία συλλογική βάση στην Ευρώπη, η συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σίγουρα η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανθεκτικότητα. Η επένδυση στην ε, ανθεκτικότητα είναι πολύ πιο σημαντική για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε κρίση. Γι' αυτό θα συνεργαστώ με τον Επίτροπο Μίμικα, που είναι υπεύθυνος για θέματα ανάπτυξης. Πέμπτον, χρειαζόμαστε μία κοινή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε την κρίση έμπολα. Εργαζόμαστε στην Επιτροπή επί του θέματος μέσω του Κέντρου Συντονισμού Επίγουσας Ανταπόκρισης, ERCC, που συνδέεται με τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς εταίρους μέσα στα πλαίσια των μεγάλων χορηγών ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειλικρινά όμως τα αποτελέσματα δεν έχουν φτάσει. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Έκτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε προστατεύοντας τους Ευρωπαίους πολίτες. Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας πολιτικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πλέον αξιόπιστη και προβλέψιμη καθώς και αποτελεσματική απάντηση στις μεγάλες καταστροφές. Τέλος, σε σχέση με την συνεκτική προσέγγιση, θα συνεχίσω το έργο της προκατόχου μου. Είμαστε εντός αλλά εκτός. Γι' αυτό, εάν διοριστώ, θα συνεργαστώ με την ύπατη εκπρόσωπο και άλλους επιτρόπους για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τη ρίζα της κακοδαιμονίας, κακοδαιμονίας και να μπορέσουν οι χώρες να επανέλθουν στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα συνεχίσω να διασφαλίζω την, τις πραγματικές αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας να έχουν πρόσβαση στα θύματα και να μπορέσουν να τα βοηθήσουν. Τους το χρωστάμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες βρέθηκα σε βαθιά νερά εκπαίδευσης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο ε, περιέχει πολλά θέματα επίγουσας ε, βοήθειας και αντιμετώπισης καταστάσεων κατεπήγοντος. Εάν ε, όμως επειδή μαθαίνω πολύ γρήγορα, σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι νύχθη μερών για, τα, για να κατανοήσω καλύτερα τα θέματα αυτά. Και θα έρχομαι πολύ συχνά στην Επιτροπή σας για να συζητώ αυτά τα ζητήματα μαζί σας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη για την εξαιρετική αυτή εισαγωγή και τώρα θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις από πλευράς των πολιτικών ομάδων, ξεκινώντας με τον κύριο Στήρο από πλευράς της ε, ομάδας του ΕΛΚ. Ένα λεπτό και μετά follow-up. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στο, στο ξέσπασμα της ε, έμπολα και πολύ σωστά το θέσατε μεταξύ των προτεραιοτήτων της εργασίας του Επιτρόπου. Στη συζήτηση που έγινε, για παράδειγμα στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, υπήρξαν εκτιμήσεις 20.000 προσβεβλημένων μέχρι τα τέλη του χρόνου. Αυτό πριν από κάποιες εβδομάδες, στο Στρασβούργο. Αυτή ήταν η εκτίμηση. Και τώρα έχουμε από το Κέντρο για την Πρόληψη των Νόσων μια εκτίμηση για 4,4 εκατομμύρια προσβεβλημένους μέχρι τον Γενάρη, αν δεν αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά της διεθνούς κοινότητας. Μας είπατε ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι πώς αξιολογείτε, αν θέλετε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες, τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και πιο συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο. Allow me to continue in my mother tongue. Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η διεθνής κοινότητα έχει καθυστερήσει. Υποτίμησε τον κίνδυνο του έμπολα. Μόνο έτσι θα ξεκινήσουμε σωστά. Είναι γνωστή η διατύπωση του επιδημιολόγου Προέδρου της World Bank που είναι και ειδικό ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι μια θέση ειδικού πρέπει να δράσουμε σύντομα. Πιστεύω ότι η επιστολή που στείλατε ήδη ως κομίτη βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι, χρειάζεται άμεσα, και μιλώ τώρα και με την ιατρική μου ιδιότητα, χρειάζεται άμεσα, χρειάζονται άμεσα γιατροί επιτόπου. Χρειάζεται νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται να ασκηθούν νοσοκομεία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Όχι αύριο μεθαύριο. Διότι όντω, εάν περάσει η ασθένεια σε αστικού πληθυσμού, δεν μπορεί να τη μαζέψει κανεί. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε συντονισμένα. Και ο συντονισμός σημαίνει ότι πρέπει όλοι οι international partners, οι διεθνείς εταίροι να βρεθούν κοντά. Τα member states να δράσουν κατά τρόπο που να είναι αποτελεσματικός. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Η επερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Μπορείτε να εντοπίσετε τώρα, σε περίπτωση που διοριστείτε, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα βήματα που θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε το ξέσπασμα της επιδημίας έμπολα ως νέος επίτροπος. Εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θεωρώ ότι η πολιτική μου συνείδηση και η ιατρική μου ιδιότητα μου επιβάλλουν να είμαι παρόν στις πληγίζες περιοχές ως την πρώτη μου ενέργεια, ως το πρώτο μου ταξίδι. Εκεί θα δω επιτόπου την κατάσταση για να μπορέσω όντως να συντονίσω και να διαμορφώσω η ανάποψη. Εκεί μπροστά στις πληγίζες περιοχές τους ασθενείς θα ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να μπορέσω να διαμορφώσω συγκεκριμένο σχέδιο και για τη συνεργασία και τον συντονισμό αλλά και επί του εδάφους. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο ταξίδι. Αυτή είναι η δέσμευσή μου, αγαπητέ συνάδελφε, και θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητε γιατί στέλνουμε το μήνυμα κιόλα και σε συναδέλφους γιατρούς αλλά και σε άλλους, ναι, ότι πρέπει να πάμε εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι του κυρίου Λίτς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ συναισθηματική και έντονη εισαγωγή που κάνατε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ε, ανθρωπιστικής κρίσης τώρα. Συμφωνώ λοιπόν με την εισαγωγή που κάνατε. Έχω μία ερώτηση να σας απευθύνω για την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον τρέχον κανονισμό του Συμβουλίου. Ο 1275 του 96 από το 1996 χρήζει αναθεώρησης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανθρωπιστικές ανάγκες και να ενημερωθεί σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία που εισήγαγε η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει αναβληθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία από πλευρά τη ε, Επιτροπή. Οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε έχουν πολλέ φορέ καλέσει για να αναθεωρηθεί ο κανονισμό αυτό, προκειμένου να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα ε, της αντιμετώπιση των κρίσεων, όπως υποδείξατε και εσείς στην αρχή. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να γίνει τέτοια αναθεώρηση πριν τα τέλη του 2016 και αν όχι, γιατί όχι. Και αν ναι, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης, ποια θα πρέπει να είναι τα στοιχεία της αναθεώρησης. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έχετε απόλυτο δίκιο και από ό,τι έχω ενημερωθεί, όντω υπήρξε και μια δέσμευση για αναθεώρηση του regulation. Έχω μια άποψη στη ζωή και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σα. Πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα στατικό. Όλα αναθεωρούνται και πρέπει να είμαστε έτοιμοι στη βάση των νέων συνθηκών και αναγκών να αναθεωρούμε πράγματα. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι στις αναθεωρήσεις. Στη βάση του αξιώματος ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν λάθη. Όμως πιστεύω ότι εάν είναι έντονη η θέση από ένα μεγάλο κόμμα όπως οι σοσιαλιστές δημοκράτες θα πρέπει όντως να ανοίξει ένας διάλογος και να το κουβεντιάσουμε, να δούμε εις βάθος πού μπορεί, να γίνουν αναθεωρήσεις και αν προκύψει κοινή θέση και κοινή στάση, σε αυτή την περίπτωση, ναι, να δούμε πώς θα το προωθήσουμε. Ξέρετε βέβαια ότι απτείται του κολεγίου η απόφαση αυτή. Εγώ τουλάχιστον αυτό που μπορώ να σας πω, παρόλο που επαναλαμβάνω υπάρχει η περίπτωση να μην χρειάζεται γιατί φαίνεται ότι δουλεύει, Είμαι έτοιμος στον επόμενο χρόνο να κάνουμε αυτή τη διαβούλευση μέσα στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής και να δούμε όλα τα κόμματα εάν μπορούμε όντως να προωθήσουμε αναθεώρηση. Εάν προκύψει ότι δουλεύει ο κανονισμός, να παραμείνουμε ως έχει. ευχαριστώ. Μία επερώτηση αναφερθήκατε στην κατάσταση σε ό,τι αφορά το ξέσπασμα έμπολα. Ο συντονισμό και στο Ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων φορέων είναι κάτι το απαραίτητο για αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να φτάσει στου ε, ανθρώπου που τη χρειάζονται. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. Και πρόσφατα συναντηθήκαμε με τον Ευρωπαίο πρέσβη στο Ιράκ που έδωσε σχετική αναφορά στο Κοινοβούλιο και μας Ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού με διεθνεί οργανισμού, όπω ο ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων επιτόπου και σε ό,τι αφορά την επιδημία έμπολα. Η κατάσταση θα πρέπει να επιληθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι βήματα συγκεκριμένα προτείνεται για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και με τους άλλους διεθνείς φορείς. Το θέμα του συντονισμού είναι το κύριο υπόβαθρο για να έχει αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μία πρακτική. Ειδικά στην περίπτωση του έμπολα, δίχως συντονισμό, όλα είναι στον αέρα, είναι μετέωρα. Με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι ε, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους. Έχω ήδη έρθει σε επαφή με κάποιες σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο των Ηνωμένων Εθνών την κυρία Βαλεριάμος από την Ότσα, τον κύριο Κουτέρες από, είπα το εκπρόσωπο για τους πρόσφυγες και είμαι σε μια επαφή μαζί τους και αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας θα μπορέσω αυτή την επαφή να τη συνεχίσω έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ πρακτικό επίπεδο αποτελεσματικοί. Πιστεύω ότι είναι εκ των ουκάνευ, είναι συνεκβανών η συνεργασία των, εταίρων, των διεθνών εταίρων με τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Δράσης. Αυτό είναι υπόβαθρο για να χτίσουμε το μέλλον. Ειδικά στον έμπολα, είπα και πριν ότι υποτιμήθηκε, υπάρχουν σήμερα νέα δεδομένα, εγρήγορση, κινητοποίηση από πλευρά διεθνού κοινότητα και πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο ε, από τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Πίτροπε, το 2016 θα γίνει παγκόσμια διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη για την ανθρωπιστική βοήθεια και πιστεύω ότι θα δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα τη μάστιγα του AIDS. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει να ορίσουμε στόχους για την περίοδο μετά το 2016 για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πώς θα ορίσετε τους ευρωπαϊκούς ε, στόχους. Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διάσκεψη κορυφής. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί όντως η διάσκεψη κορυφής του 16 στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Για τρεις λόγους. Το πρώτο δεν είναι διακυβερνητική, δεν είναι intergovernmental διάσκεψη. Θα είναι όλοι οι παράγοντες της διεθνούς ανθρωπιστικής κοινότητας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους. Ο ένας είναι innovation, ο δεύτερο είναι αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα τη ανθρωπιστική δράση, vulnerability και έχει σχέση ακόμη και με το γεγονό ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανθρώπων στην κρίση, το access, την πρόσβαση. Εσεί θέσατε ακόμα ένα θέμα, το θέμα του AIDS, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο. Λοιπόν, εκεί σε αυτή τη διάσκεψη θα υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξουν τα θέματα. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να πάει με μια πολύ σημαντική προετοιμασία. Γι' αυτό έχουμε πρώτη άσκεψη στο Βουκουρέστι το 2015 και πιστεύω ότι πρέπει ο Επίτροπος, εάν με τιμήσετε με την έγκρισή σας, μαζί με την Επιτροπή, την ΤΕΒΕ, θα πολλαπλασιάζονται και πρέπει να ανταποκριθούμε με Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε δια της ευελιξίας, η οποία δεν επαρκεί σε αυτή την ε, περίπτωση κρίσεων. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα αποθεματικά μας, το αποθεματικό μας και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι το παράλογο το οποίο εγγράφεται στο σύστημά μας στην ανισορροπία μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Όταν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε και τους τελευταίους πόρους και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, τότε βρισκόμαστε χωρίς μέσα για τις μελλοντικές προκλήσεις των ανθρωπιστικών κρίσεων. Εδώ πρόκειται για ένα συστηματικό λάθος ή μία έλλειψη. Πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, την έκρηθμη κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο στον τρόπο που περιγράφετε την κατάσταση και ξέρω ότι είστε άνθρωπος που ασχολείστε χρόνια με αυτά τα θέματα στη συγκεκριμένη Επιτροπή επειδή είμαι μέλος της budget ως Ευρωβουλευτής και αυτό το δίμηνο έχω αποκτήσει κάποια μικρή εμπειρία γύρω από το θέμα και σήμερα έχουν περάσει σημαντικά θέματα που αφορούν την ΤΕΒΕ και τον προϋπολογισμό. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει από κοινού να πείσουμε για την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής δράσης ότι δεν είναι μια συνηθισμένη δράση. Γι' αυτό θα πρέπει να τύχει μια ειδική μεταχείριση στα θέματα προπολογισμού. Και πολύ σωστά είπετε, θα πρέπει να έρθει η στιγμή που τα payment και τα commitments να εξισωθούν. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αναγνωρίζω ότι είναι γενικότερο πρόβλημα του προπολογισμού στην Ένωση. Όμω, για μα, στην ανθρωπιστική δράση πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο. Και έχουμε επιχειρήματα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί τα επιχειρήματα που έχουμε για την ιδιαιτερότητα. Εάν καταφέρουμε μέχρι το 2016 να φτάσουμε σε αυτή την εξίσωση, χρησιμοποιώντας και λεφτά από το αποθεματικό, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε όντως τη δυνατότητα η ανθρωπιστική δράση να μην μειωθεί παρόλο που ανεβαίνουν οι ανάγκες. Θα έλεγα όμως ένα επόμενο βήμα είναι ότι πρέπει να ψάξουμε για νέους χορηγούς. Γι' αυτό ανέφερα πριν την αξία της Κωνσταντινούπολης ως του συμβολικού σημείου του Σάμιτ. Άρα, αν μπορώ να ερμηνεύσω όσα προείπατε, θα περιμένετε την ενδιάμεση αναθεώρηση έτσι ώστε να δείτε ποιο μέρος του προϋπολογισμού θα ε, επιδοθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένα κατά παρέκκληση καθεστώς που να διέπει την ανθρωπιστική δράση. Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015, να επιμείνουμε στη θέση της ιδιαιτερότητας. Και θεωρώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο στα πλαίσια των συζητήσεων να τεθεί όντω το ζήτημα της ιδιαιτερότητας με πολύ έντονο και άμεσο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι η μόνη δράση που έχει τόσο έντονο το στοιχείο του επίγοντος. Ότι δεν μπορεί να τα προβλέψεις όλα. Και αυτό ακριβώς επιβάλλει αυτή τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στο αποθεματικό emergency, αλλά την ίδια στιγμή να έχει τη δυνατότητα τα payments και τα commitments να είναι εξισωμένα. Εξάλλου όλοι ξέρουν ότι οι χορηγίες προς τα NGOs δυστυχώς δεν μπορούν να αργήσουν, διότι τα NGOs δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τράπεζες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν αυτά τα λεφτά την ώρα που χρειάζονται. Γιατί μόνο έτσι θα σώσει ζωέ. Έτσι θα μειώσει τον πόνο και το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Χρυσόγονος, ο οποίος κάθεται πίσω σας, κύριε Επίτροπε, και θα σας μιλήσει μάλλον στα ελληνικά, από την ΚΟΕ. Ε, ε, ε, κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, στο παρελθόν υπήρξαν επανειλημμένα σοβαρές καταγγελίες για κρούσματα κακοδιαχείρισης αν μη και διαφθοράς, σε σχέση με την υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ε, χώρες του τρίτου κόσμου, παραδείγματος χάρη στη Σομαλία. Εφόσον επιβεβαιωθείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε εάν ανακύψει μια παρόμοια περίπτωση στη διάρκεια της θητείας σας ως Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Όντως είναι μέρος της ζωής δυστυχώς και η διαφθορά και η απάτη. Και υπήρξαν κάποια κρούσματα και από ό,τι πληροφορήθηκα έγιναν παρεμβάσεις σε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο η ενημέρωσή μου μου λέει ότι ναι, υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, υπάρχει έλεγχος από εμπειρογνώμονες και φτάνουμε στο Court of Auditors. Υπάρχει δηλαδή ένας έλεγχος και φαίνεται από την αξιολόγηση ότι όντως είναι αποτελεσματικός. Και μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη τουλάχιστον με βάση την αξιολόγηση που γίνεται ότι είναι πολύ ψηλά στην κλίμακα της, του, της διαβάθμισης όλων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στην ΕΚΟ. Όμως δεν είμαστε αφελείς. Ξέρουμε ότι <laughs> υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαφθορά και απάτη. Πιστεύω ότι πρέπει και μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, γνωρίζοντα καλύτερα και σε περισσότερη λεπτομέρεια το όλο σύστημα, μαζί με ειδικού ανθρώπου να το βελτιώσω όσο είναι δυνατόν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ανα πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Εκεί θα πρέπει βέβαια να επιδειχθεί πολιτική βούληση. Να αντιδράσουμε με ένα καθαρά πολιτικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης πολιτικής βούλησης και της άτεγκτης στάσης την οποία μας εξαγγέλλεται σε ηθικά ζητήματα θα ήσασταν διατεθειμένος να φτάσετε μέχρι και στο σημείο ε, διακοπής ε, ενός προγράμματος ή αντικατά, άμεσης αντικατάστασης των υπευθύνων διαχείρισής του εφόσον συντρέχει περίπτωση. Σαφέστατα κύριε συνάδελφε. Δεν, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα πρέπει ναι να είμαστε αμήλικτοι στα θέματα διαφθοράς και απάτης. Δεν πρέπει τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων να βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να προκύψουν απάτες και να μην πάνε εκεί που πρέπει ειδικά τα, τα λεφτά της ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι ιερά. Είναι λεφτά που πάνε για να σώσουν ζωές, είναι λεφτά που πάνε για να φάνε παιδιά, είναι λεφτά που πάνε για να μην χάσει μια γενιά το μέλλον της. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αμήλικτοι και σε αυτά δεν πρέπει να σηκώνουμε κουβέντα. Όπως λέμε στα ελληνικά, όπως καλά ξέρετε. Λοιπόν, δεσμεύομαι γιατί το θεωρώ δέσμευση αυτό. Όταν προκύψει τέτοιο θέμα το πρόγραμμα πρέπει να σταματά και να ξεκινούν όλες οι διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει πάρα πολύ αυστηρές. Έχω την εντύπωση από την ενημέρωση που έτυχα, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, 15-17 μέρες, ότι έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα και έχει επιδειχθεί μια τέτοια αμήλικτη στάση. Thank Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Χάουταλα από την ομάδα των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι βέβαιη ότι όλοι εκτιμούμε το όραμα που μας παρουσιάσατε. Μιλήσατε για το ότι θέλετε να πολεμήσετε για τους πιο ευάλωτους. Θέλετε να είσαστε η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω μια ερώτηση. Πολλές μειονότητες υποφέρουν πιο πολύ από τι οι άλλοι από τις ανθρωπιστικές κρίσεις. Για παράδειγμα, οι ανάπηροι, τα ανάπηρα παιδιά, φυσικά και οι γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες συχνά ανήκουν, θεωρείτε ότι ανήκουν στην ε, πλειονότητα. Πώς λοιπόν μπορείτε στην πράξη να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες των πιο ευάλωτων, των ανάπηρων, των γυναικών, των παιδιών. Και έχετε οποιαδήποτε ιδέα για το πώς η ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να αφιερωθεί ειδικά σε αυτές τις ε, ευάλωτες ομάδες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις υγειονομικές ε, καταστάσεις για άτομα με αναπηρία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και την πρόληψη της σεξουαλικής ε, παρενόχλησης των γυναικών. Ποιες θα ήταν οι βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε για την ευαισθησία ακριβώς για αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Νομίζω ότι ο άνθρωπος καταξιώνεται όταν ακριβώς αντιμετωπίζει τις ευάλωτες ομάδες με την διαφορετικότητα που τους πρέπει. Αλλιώς η ζωή είναι ισοπεδωτική και αποκτά και κοινικό χαρακτήρα. Κάποιοι πρέπει να τη χάνουν όντω προνομιακή μεταχείριση. Και αυτέ είναι οι ευάλωτε ομάδε. Ειδικά τα άτομα, όπω είπατε, με κινητικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλα. Η οποιαδηποτε αλλη η ενημερωση που έχω μέχρι τώρα, δεν λέω ότι είμαι ειδικό στο θέμα και ίσω θα πρέπει να εμβαθύνω περισσότερο στο θέμα και να σα δώσω πιο συγκεκριμένε απαντήσει. Αλλά η ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα είναι ναι. Στου δείχτε και στα κριτήρια που προσφέρεται ανθρωπιστική βοήθεια μέσω εξειδικευμένων ε, ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα θέματα γυναικών, παιδιών, σεξουαλικής βίας παρενόχλησης και τα ζητήματα που αφορούν σε άτομα με ειδικέ ανάγκες. Εάν έχουμε δυνατότητα θα πρέπει να το επεκτείνουμε και έχετε δίκιο. Εκεί ακριβώς θα αναδειχθεί η βασική αξία τη ανθρωπιστική δράση που είναι ο ανθρωπισμό. Η μία από τι βασικέ μα αρχέ. Ο ανθρωπισμό δεν είναι θεωρητική έννοια. Πρέπει να έχει πρακτική αξία. Και στην αντιμετώπιση των ευάλωτων ομάδων πρέπει να έχει πρακτική αξία μέσω δικτών και κριτηρίων. Ναι, έχω και μία επερώτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι εκατομμύρια παιδιά μένουν σε εγκαταστάσεις προσφυγικές επί μακρά περίοδο, 20 έτη. Στην Κένια, για παράδειγμα, υπάρχουν άτομα τα οποία 20 χρόνια ζουν σε τέτοιες εγκαταστάσεις μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης και στην ε, Ιορδανία σε ένα μικρό χωριό το οποίο ε, διαχειρίζεται, το διαχειρίζονται σαν ε, μια μικρή πόλη ουσιαστικά. Στην πρώτη λοιπόν σύνοδο ανθρωπιστικής κρίσης θα μπορούσατε να δώσετε κάποια ελπίδα στα άτομα που ζουν σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Ένα σχέδιο για τους πρόσφυγες λοιπόν θα μπορούσατε να το προωθήσετε. όντως όπως το περιγράφεται είναι μια μεγάλη πρόκληση την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε εις βάθος και να βρούμε τους πρακτικούς τρόπους της προώθησης αυτών των θεμάτων που δυστυχώς είναι τόσα χρόνια άλυτα. Γιατί μετά χάνουμε γενιές ολόκληρες και αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα και δυστυχώς στη Συρία. Ξέρετε τι συμβαίνει επί του εδάφους. Έξι εκατομμύρια παιδιά ενδεχομένως έχουν ήδη υποστεί τις πληγές και τα τραύματα του πολέμου. Στην Κένια, στο Νότιο Σουδάν, στο Κόγκο υπάρχει εκτός που το πρόβλημα το γνωστό του υποσυτισμού που προσφέρουμε φαγητό υπάρχουν και τα ψυχικά τραύματα, υπάρχουν και η έλλειψη προοπτικών. Ένα παιδί αν δεν έχει προοπτικές για να συνεχίσει τη ζωή του ουσιαστικά το καταδυναστεύει, βιώνει τα τραύματα αυτά και δεν μπορεί να συνεχίσει παρακάτω. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα θέματα που ενδεχομένως στην Κωνσταντινούπολη να τα αναδείξουμε ως μέρος της κοινή μας ευρωπαϊκής θέσης. Thank you. Mr. Ο κύριος Κοράου από την Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας κύριε Επίτροπε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, την μεγάλη καταστροφή στον ε, κόλπο του Μεξικού καθώς και την καταστροφή της ε, Φουκουσίμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δυνατές χώρες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστροφές. Αυτό σημαίνει ότι τα ενεργειακά μας πρότυπα δεν είναι πάντα σωστά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά, ε, υπάρχουν πολλά δηληστήρια, καθώς και πυρηνικές μονάδες, που θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες. Εάν λοιπόν μετά από τρεις μήνες υποστούμε μία φυσική καταστροφή σαν αυτή της Φουκουσίμα ή του κόλπου του Μεξικού, θεωρείτε ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαίοι και αν ναι Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μας εισαγάγει ουσιαστικά στη δεύτερη διάσταση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Δράσης που είναι η πολιτική προστασία. Στη Φουκοσίμα, που έχετε δίκιο μια μεγάλη χώρα όπως η Ιαπωνία, ζήτησε βοήθεια και η Ευρώπη ήταν εκεί να βοηθήσει. Έχουμε πάρει πολλά διδάγματα για το θέμα των πολυτομεακών καταστροφών που προέρχονται από φυσικά φαινόμενα. Λέω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας ο οποίος βασίζεται και στη λογική της προετοιμασίας σχεδίων και του prevention. Θέλει οπωσδήποτε ετοιμότητα. Και υπάρχει μια πολύ σωστή σχέση, εξελίσσεται μια πολύ σωστή σχέση μεταξύ του ίδιου του μηχανισμού και των κρατών μελών στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι ένα καλό παράδειγμα που μου δίνει τουλάχιστον εμένα ελπίδε είναι αυτό που ανέφερα και στο opening statement μου για το θέμα τη Βοσνία. Όπου τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τι πλήμμυρε του 2001. Και εκεί ήταν μια πολυτομιακή. Είναι διάφορε εμπειρίε, έχουν σχέση και με πυρηνικά ατυχήματα και όλα, τα οποία θα πρέπει όντω να κωδικοποιήσουμε περισσότερο και να είμαστε προληπτικοί. Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία. Χρειάζονται πολλά να γίνουν στο επίπεδο τη πρόληψη και ο μηχανισμό πολιτική προστασία προσφέρεται ω υπόβαθρο να χτιστεί αυτή η πρόληψη. Στη Σικελία υπάρχουν τρεις μονάδες υψηλού κινδύνου και στο δηληστήριο του Μιράτσο στην Σικελία ε, ξέσπασε φωτιά και ήδη ζούμε μία κατάσταση που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Θεωρείτε ότι η διαχείριση αυτών των κινδύνων θα πρέπει να περάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να μην αντιμετωπίζεται εθνικά ή τοπικά. δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στη Σικελία. Το ομολογώ. Αλλά ξέροντας και ενημερωνόμενος για την μηχανισμό πολιτικής προστασίας, σας λέω ναι, από τη στιγμή που ζητηθεί βοήθεια από ένα κράτος μέλος, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι έτοιμο να τον παράσχει. Και μάλιστα να ζητήσει συνδρομή και άλλων κρατών μελών. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές σε πυρκαγιές στην Νότια Ευρώπη, ακόμα και διασυνοριακά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι και εντός των ευρωπαϊκών συνόρων και εκτός. Που σημαίνει είναι θέμα να υπάρξει αίτημα για να υπάρξει βοήθεια. Πιστεύω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά γύρω από αυτό το θέμα. Έχουμε το κέντρο, το ERCC, το κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο από ό,τι είδα και με κάνει περήφανος Ευρωπαίο, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση και να προλάβουμε τραγικές εξελίξεις πιστεύω ότι είναι θέμα έτοιμα του κράτους μέλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θέμα πιο τοπικό, δεν το γνωρίζω. Μπορώ όμω σε άλλο επίπεδο να το κουβεντιάσουμε αφού μάθω λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος των ομιλητών και τώρα έχουμε δύο ομιλητές από τις επιτροπές που μας επισκέπτονται. Ο κύριος είναι ο κύριος Πρέντας από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ. Το χαρτοφυλάκιό σας είναι πολύ σημαντικό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ανθρωπιστικής βοήθειας και επειδή πρόκειται για μια ουσιώδη δραστηριότητα της Ένωσης, είμαι πεπισμένος ότι διαθέτεται όλες τις αρμοδιότητες για να φέρετε εις πέρας την αποστολή σας. Από πλευράς ΑΦΕΤ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα συνεργαστείτε με την ύπατη εκπρόσωπο έτσι ώστε να μην υπάρξει αποσύνδεση με την εξωταρική πολιτική και την ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στα πλαίσια της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανθρωπιάς, όπως είπατε. Θα ήθελα να μας μιλήσετε και για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ξέρετε πολύ καλά ότι χορηγήσαμε μεγάλη βοήθεια, αλλά είναι δύσκολο να μπούμε στις ζώνες σύραξης. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έχετε απόλυτο δίκαιο ότι πρέπει ο συντονισμός, η συνεργασία στο επίπεδο του project team, όπως τα όρισε ο πρόεδρος Επιτροπής κύριο Γιούγκερ, θα πρέπει να είναι συστηματική και πρακτική. Γι' αυτό και έχει αξία το project team των external affairs του οποίου συντονίστρια είναι η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη ως αντιπρόεδρος και high representative. Σε ό,τι αφορά τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Δράσης. Είπα και στην αρχική μου παρέμβαση ότι θα συνεχίσω στη γραμμή της κυρίας Γεωργίευα, η οποία απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Επιμένουμε στο in but out. Ναι, θα παρέχουμε τις πληροφορίες, την ανάλυση εκτιμήσεων, δεδομένα που μαζεύουμε από το εκατοτόπους γραφεία τους εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να είμαστε μέρος της συλλογικής δουλειάς του Project Team για αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων και χρειάζονται πολιτικές λύσεις, το ξέρουμε όλοι. Είναι γνωστή και η διατύπωση του Ιάπωνα ανθρωπιστή ότι δυστυχώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν ανθρωπιστικές λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα. Χρειάζονται πολιτικές λύσεις για να έχουμε τελική κατάληξη. Απλώς οι ανθρωπιστικές λύσεις είναι για να ανακουφίσουν. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, ναι, στο project team θα έχουμε σημαντικό ρόλο στη συζήτηση της πολιτικής. Αλλά την ίδια στιγμή, και έχετε δίκιο, θα πρέπει να κρατήσουμε τις τέσσερις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής δράσης. Εάν δεν τις κρατήσουμε, θα σταματήσουμε να έχουμε πρόσβαση, access, εις αυτούς που έχουν ανάγκη στα θύματα. Γι' αυτό πάση θυσία θα είμαστε in, but out για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κρατήσουμε το κύρος και τις αξιοπιστίες ανθρωπιστικής δράσης. Σας ευχαριστώ κυρία Γκαρτίνη τώρα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την πολιτική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σταθούμε στο νέο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ήμουνα εισηγήτρια επί του θέματος και υπήρχε συμπαγής στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε με βάση αυτό το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες δράσεις θα αναλάβετε έτσι ώστε να δράσει αποτελεσματικά ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και πώς μπορεί να γίνει συντονισμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Επίτροπης μέσα στα πλαίσια των κρατών μελών και της εθνικής πολιτικής προστασίας και των κρατών που συμμετέχουν στο μηχανισμό σε σχέση με τον επιμερισμό ε, μέσων και το voluntary pool. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να είναι σημείο εκκίνησης για το συντονισμό αυτού του μηχανισμού. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή εργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακρίνω ότι γνωρίζετε εις βάθος το θέμα. Και θα σας πω πολύ απλά ότι στα πλήστα που είπετε συμφωνώ. Και όντως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι ο μηχανισμός που συνδέει τα κράτη-μέλη με την Επιτροπή στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Συντονίζει ουσιαστικά μέσω του κέντρου του ERCC, συντονίζει ακριβώς τα κράτη-μέλη πώς θα βοηθήσει το ένα το άλλο. Για να έχουμε συλλογική δουλειά. Και θα επαναλάβω το παράδειγμα της Βοσνίας. Τώρα, ότι μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις, οπωσδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα στη λογική της πρόληψης να ετοιμαστούν σχέδια, να υπάρχει η δυνατότητα του buffer όπως λέμε, έτσι ώστε εάν προκύψει ανάγκη σε μια άλλη χώρα να βοηθηθεί από την συλλογική δουλειά των υπολείπων χωρών και αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προγράμματα που για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως σχέδιο που εμπίπτει στα πλαίσια του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δεσμεύει τις χώρες. Σε ό,τι αφορά το, εθελοντικό, έχετε δίκιο ότι το εθελοντικό προσφέρει δυνατότητες. Θα πρέπει να το επεκτείνουμε και να του δώσουμε μια περισσότερη πολιτική δύναμη θα έλεγα στο βαθμό που θα αποκτήσει ένα συγκεκριμένο ρόλο στον όλο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που αποδεικνύεται στην πράξη, που βοηθά και διασυνοριακά. Δεν είναι μόνο 28 χώρες, είναι και η Νορβηγία και η Ισλανδία και έκανε αίτηση και, το Μοντενέκρο και το Ιφυρόμ και αυτό αποδεικνύει ότι και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης θέλουν να ενταχθούν στο μηχανισμό. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στις πολιτικές ομάδες. Πρώτος ομιλητής είναι η κ. Πόγκα. Αντιπρόεδρος και είναι πίσω σας. Κύριε Επίτροπε, τα μέτρα πρόληψης και μείωσης κινδύνων έχουν μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σειράξεις αλλά και τις φυσικές καταστροφές που είναι όλο ένα και περισσότερες. Ποια στρατηγική θα θέσετε σε εφαρμογή για να μειώσετε την ευαλωτότητα των ε, ε, τοπικών κοινοτήτων. Οι συνέργειες αυτές θα πρέπει να προωθηθούν μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης και πώς θα πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την μαγική λέξη ότι ναι, για να μπορέσουν να αποκτήσουν νόημα όλες οι πολιτικές μείωσης κινδύνων και να προχωρήσουμε στο resilience χρειαζόμαστε την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία του κυρίου Μίμητσα. Γι' αυτό δεν μπορεί να μην λειτουργήσουμε συμπληρωματικά. Η ανθρωπιστική δράση ανακουφίζει, η ανθρωπιστική δράση δρά τη στιγμή που υπάρχουν οι ανάγκες αλλά μετά αρχίζει η δράση της ανάπτυξης. Το λεγόμενο LRT ανακούφιση, αποκατάσταση και μετά ανάπτυξη. Αυτά τα τρία πρέπει να συνδέονται. Και όσο πιο καλά συνδέονται, τόσο πιο καλά αποτελέσματα έχουμε. Ήδη έχω κάνει μία συνάντηση με τον συνάδελφο τον κύριο Μίμητσα, συζητήσαμε ακριβώ πάνω σε αυτό το θέμα, ειδικά στο επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων. Εκεί είναι η αξία τη αποκατάσταση και ανάπτυξη. Νομίζω έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στο Σαχέλ το Αζίρ, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιούμε ως εμπειρία για να μπορούμε με αυτά τα διδάγματα που έρχονται από το Αζίρ να επεκτείνουμε και τις πρακτικές μας και τις πολιτικές μας. Υπάρχει ανάλογο παράδειγμα βέβαια και στο κέρα της Αφρικής, το ΣΕΑ. Λοιπόν, ε, έχετε δίκιο ότι πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περαιτέρω τη στρατηγική, θα πρέπει να δούμε τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινότητες. Αυτό θα βοηθηθούμε από τα τοπικά NGO που θα τα βοηθήσουμε να έρθουν σε συνεργασία με τα NGOs τα οποία είναι γνωστό ότι ε, χορηγούνται από εμά, τη χάνουν χορηγία από εμά και αυτό θα δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για να μπούμε στο resilience building. Σα Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι, είναι ο κ. Γκανσαλάμ από τους Σοσιαστές και Δημοκράτες. Κύριε Στυλιανίδη, δύο ερωτήσει σε μία. Καταρχήν, στα πλαίσια του χαρτοφυλοκίου σας θα πρέπει να διαχειριστείτε και κρίσεις. Αυτό αφορά τη μετανάστευση, την κινητικότητα και τους πρόσφυγες. Αυτό γίνεται στις όμορες με την Ένωση περιοχές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο θα τηρηθούν τα δικαιώματα των προσφύγων στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής με τον αρμόδιο επίτροπο επιθεμάτων μετανάστευσης. Επίσης, στην παρέμβασή σας μιλήσατε για πρόληψη. Πρέπει να δράσουμε σήμερα και όχι αύριο δεν πρέπει να δράσουμε too little ή too late. Και υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να συνεργαστείτε με την κυρία Γεωργίεβα, η οποία τώρα θα ασχοληθεί με τους προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο 50 εκατομμύρια για μια κρίση όπως αυτή της Συρίας με εκατομμύρια πρόσφυγες. Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε δίκιο ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις στην περιφέρεια της Ευρώπης έχουν φτάσει στην κορύφωσή τους και έχουμε πρόσφυγες που δημιουργούν μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Συρία. Στην Τουρκία τρεις μέρες πέρασαν 138.000 πρόσφυγες. Αυτό είναι τρομακτικό σαν αριθμός όταν το σκεφτούμε. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει αυτή την κατάσταση και έχει απόλυτο δίκιο. Αρμόδιος Επίτροπος για μετανάστευση υπάρχει και ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιούγκερ, γι' αυτό όρισε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα θέματα μετανάστευσης. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό. Και ο ρόλος του δικός μου και η συνεργασία με τον κύριο Αβραμόπουλο είναι δεδομένη. Και στα πλαίσια του project team, αλλά και σε κατηδίαν επαφές. Όμως ως Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δράσης, εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, αυτό που θα κάνω πρώτιστα είναι ακριβώς πώς θα αντιμετωπίζω τα ανθρωπιστικά προβλήματα αυτών των ανθρώπων εκεί που είναι. Στα καταλήμματα, το πώς τα παιδιά δεν θα χάσουν τη σχέση τους με την παιδεία, το education, στο πώς θα φάνε, στο πώς θα έχουν πόσιμο νερό, υγιεινή αποχέτευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενδεχομένως να δημιουργήσει και αποσυμπίεση κάπου το μεταναστευτικό ρευμάτων. Ενδεχομένω λέω. πάση περιπτώσει, σημασία έχει ως Επίτροπο Ανθρωπιστική Βοήθεια, διατηρώντα την αξιοπιστία σε επίπεδο ανεξαρτησία, μακριά από μένα η οποιαδήποτε λογική η ανθρωπιστική δράση να γίνει εργαλείο πολιτικής διαχείρισης, τότε χάνει το νόημά της, χάνει τη σημασία της τότε δεν θα κάνει τη δουλειά της και γι' αυτό θα μπορεί να δράσει αποτελεσματικά ακριβώς στο επίπεδο που είπατε εσείς. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Σουλούκη από πλευρά των Ευρωπαίων Συντηρητικών και των Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά τις ε, απειλές ε, των προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στο πρόβλημα. Υπάρχουν περιστατικά όπου δολοφονήθηκαν αυτοί που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο ε, με την παρανόηση ότι απειλούσαν. Απειλήθηκαν επίσης από τρομοκρατικές ισλαμιστικές οργανώσεις οι οποίες εν μέρη ήθελαν που προκαλέσουν και προσοχή στις ε, οργανώσεις τους. Και αυτό απειλεί λοιπόν αυτούς που παρέχουν βοήθεια. Πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση και είσαστε επί της αρχής διτεθειμένος να έχετε στρατιωτική βοήθεια για τα στρατιωτική βοήθεια και προστασία για το ανθρωπιστικό αυτό ανθρωπιστικό προσωπικό ή αρνείστε αυτή τη στρατιωτική ε, προστασία του ανθρωπιστικού προσωπικού. Αγαπητέ συνάδελφε, μου δίνετε την ευκαιρία να ξαναθυμίσω και να τιμήσουμε τα θύματα της ανθρωπιστικής δράσης και να καταδικάσουμε με αποτροπιασμό αυτούς οι οποίοι φτάσαν στα εγκλήματα. Θα πω από την ενημέρωσή μου ότι έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας, security γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία υπάρχουν ειδικά NGOs που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταρτίζουν τους εργάτες της ανθρωπιστικής δράσης, αυτούς τους ιδεολόγους, κατά τρόπο αποτελεσματικό το πώς θα μπορέσουν να αποφύγουν κακοτοπιές στον τρόπο που δρούν, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους. Αντιλαμβάνεστε όμω ότι επί του εδάφου η κατάσταση πολλέ φορέ είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα όντω που πρέπει να συζητήσουμε και αν μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη δυνατότητα ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, διότι βρισκόμαστε σε εντελώ διαφορετικέ συνθήκε. Στο θέμα το άλλο που αναφέρεται με τη στρατιωτική δράση. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Είμαι επιφυλακτικό στο θέμα τη στρατιωτική δράση σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική δράση. Πρέπει να είναι έσχατη ανάγκη για να μπούμε σε τέτοια δράση. Και να είναι έσχατη ανάγκη μόνο για να εξυπηρετήσει ανθρωπιστικούς σκοπούς και τίποτα άλλο. Αλλιώς θα χάσουμε την αξιοπιστία μας, θα χάσει ακριβώς την εικόνα ότι η ανθρωπιστική δράση είναι ουδέτερη, είναι ανεξάρτητη, είναι αμερόληπτη. Αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Η στρατιωτική δράση δεν πρέπει να είναι εργαλείο διαχείρισης ανθρωπιστική δράσης. Μετά οδηγούμαστε και γινόμαστε έρμεο της πολιτικής διαχείρισης και χάνουμε ακριβώ την ουσία της ανθρωπιστική δράσης. Θα χάσουμε το access και την πρόσβαση σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χάνουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Thank you, Mr. Michel. Ο κύριος Μισελ από τους Φιλελευθέρους. Ε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι όσα άκουσα μέχρι τώρα ε, με οδηγούν στο να ε, εφησυχάσω. Δηλαδή έχουμε, υπάρχουν εγγυήσεις και υπάρχει το αποτύπωμα ήδη στην Επιτροπή και χαίρομαι που και εσείς ε, έχετε δεχτεί αυτή, αυτές τις υποχρώσεις. Στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, πολλές φορές υπάρχει πληθώρα παραγόντων και πολλές φορές υπάρχει κακοσυντονισμός. Το 2010 είχαμε να κάνουμε με έναν κακό συντονισμό, κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, να σας ρωτήσω πώς θα συντονίσετε τους χρηματοδότες. Όπως είδαμε, στην περίπτωση της ΑΙΤΙΣ δεν υπήρξε καλός συντονισμός. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η θέση σας σε σχέση με την ορατότητα ή την έλλειψη ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα και εγώ ήμουν επίτροπος ανθρωπιστικής βοήθειας και έβλεπα στις σκηνές βοήθεια χορηγούμενη από τις ΗΠΑ και δυστυχώς εμείς δεν μπορούσαμε να εδραιώσουμε τη θέση μας. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και την ουσία της δράσης μέσα στα πλαίσια της ε, δράσης των χορηγών. Υπάρχει λοιπόν υπάρχει και μια αμφιβολία σε σχέση με τη στρατιωτική δράση. Ίσως θα πρέπει να, ε, να επεκταθείτε κάπως σε αυτό, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε πρόσβαση στα θύματα αν δεν υπάρχει στρατιωτική δράση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αυτά που λέτε έχουν ένα ειδικό βάρος διότι λέγονται από εσά. Ένα άνθρωπο με τόση μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι ναι, από ό,τι έχω ενημερωθεί, στα θέματα της IT υπήρξαν όντως προβλήματα συντονισμού. Και γι' αυτό ουσιαστικά περάσαμε στο αίτημα της λεγόμενης μεταρρυθμιστικής ατζέντα, του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου, έτσι ώστε να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά με βάση την εμπειρία της ΑΕΤΗΣ, γιατί υπήρξαν αυτά τα φαινόμενα. Έλλειψη συντονισμού, έλλειψη leadership, που οδήγησαν σε φαινόμενα που τα αναφέρεται πολύ καλά ότι δεν, δεν ήταν προ όφελο τη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ανθρωπιστικής δράσης. Βέβαια ήταν το φαινόμενο IT ήταν πάρα πολύ εκτεταμένο ως κρίση. Είχαμε όλα όσα μπορεί να φανταστεί κανείς. Χολέρα, τυφώνες, τα πάντα. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι η ατζέντα του ΟΗΕ των Ηνωμένων Εθνών που αφορά τη μεταρρύθμιση πρέπει όντως να ενισχυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να συζητήσει τις τρεις βασικές αρχές αυτής της ατζέντα. Leadership, accountability και συντονισμός. Coordination. Και έχετε δίκιο ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει σιγά σιγά να αποφύγουμε. Νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να συνεισφέρουμε πάρα πολύ. Ήδη σε μια συνομιλία που είχα με την κυρία Βαλερή Άμος τη Σότσα την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ό,τι καταλαβαίνω, είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά ελπίζω να έχω ευκαιρία μετά τα θέματα στρατιωτικής ε, εμπλοκής να τα κουβεντιάσω σε άλλη ερώτηση, γιατί τώρα έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος. Yes, you have minutes at the end as well. Έχετε πέντε λεπτά και στο τέλος, όπου μπορείτε να αναφερθείτε σε ποια θέματα θέλετε. Η κυρία Σάντσες Καλτέντε από πλευρά της ε, ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε, όπως είπατε και πριν, σε περίπτωση σύραξης και κοινωνικής ε, επίγουσας βοήθειας, οι πλέον ευάλωτοι είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, υπάρχουν παρενοχλήσεις, βιαιότητες και ούτω καθεξής. Είπατε στο πρόγραμμά σας αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα ήθελα όμως να μου μιλήσετε για τις συνέπειες. Πώς θα θίξετε το θέμα της σεξουαλικής υγείας και της αναπαραγωγικής υγείας σε περίπτωση σειράξεων και πιστεύετε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν παιδιά ε, μετά από βιοπραγία και βιασμούς. Το θέμα της σεξουαλικής και έμφυλης βίας δυστυχώς φαίνεται μέσα στην πληθώρα των κρίσεων έχει αναχθεί σε πρωτεύον θέμα στη Συρία, στο Ιράκ, σε αφρικανικές χώρες, στο Κόγκο, δυστυχώς είναι σε μεγάλη έκταση. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να είμαστε απολύτως καταδικαστικοί στα θέματα σεξουαλικής βίας. Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα με τα οποία υπάρχει ο χειρισμός τέτοιων περιπτώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να τύχουν αμέσω ιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης και πλήρους ενημέρωσης για ό,τι συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο που θέσατε, προσωπικά και ως ιατρός ασούμε υπέρ του ναυλώσιου. Γιατί πιστεύω, ναι, ότι η γυναίκα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να τύχει απόλυτης ενημέρωσης και να είναι η επιλογή δική της. Με βάση την νομοθεσία της χώρας και με βάση όλες τις πληροφορίες, ιατρικές, ψυχολογικές και άλλες. Η επιλογή πρέπει να είναι δική της. Γι' αυτό, γι αυτό, αυτό για μένα είναι στοιχειώδης σεβασμό στη γυναίκα. Νομίζω ότι είναι θέμα ηθικό να στηρίξουμε τη γυναίκα ακριβώς για να μπορέσει να αποφασίσει μόνη της. Σε ό,τι αφορά τα θέματα σεξουαλικής βίας σε παιδιά, κορίτσια και αγόρια ακόμη, νομίζω ότι εκεί το φαινόμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο πολύ πιο αποτελεσματικό που έχει σχέση με την ψυχολογική υποστήριξη. Είναι τόσο, σκληρές, τόσο σκληρά αυτά τα βιώματα που θέλει πολύ σοβαρή ψυχολογική υποστήριξη και ενδεχομένως εισαγωγή σε κλινικές για να μπορούν αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Thank Σας ευχαριστώ η κυρία Χάιμπρουκ για τους πράσινους τώρα. Οι κρίσεις κάθε είδους ε, οδηγούν και σε επιστικές κρίσεις και η αρρωγή σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο αλλά υπονομεύουν σε βάθος χρόνου μια τοπική και περιφερειακή οικονομία και ε, ουσιαστικά παραλύουν το σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ποια λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα κύριε Στυλιανίτη, θέλετε να λάβετε προκειμένου να φροντίσετε ότι η κατεπίγουσα βοήθεια σε επιστηστικές κρίσεις δεν θα επηρεάσει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και παραγωγή τροφίμων στις χώρες αυτές και να μπορούν να αναλάβουν η κάθε χώρα την ευθύνη της σε αυτές τις περιπτώσεις. έχετε δίκιο ότι υπάρχει ενδεχόμενο στην παροχή επιστημιστικής βοήθειας να δημιουργηθούν προβλήματα στην τοπική παραγωγή προϊόντων. Και γι' αυτό το πρόγραμμα Αζίρ στο Σαχέλ, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αυτό λήφθηκε πολύ σοβαρά υπόψη. Και αξιοποιείται πολύ σωστά μια νέα καινοτομία που έχει σχέση με το cash και το voucher. Σε συγκεκριμένε περιοχέ στη λογική του resilience building, έχουμε cash και vouchers που βοηθούν του τοπικού παραγωγού να πουλήσουν τα προϊόντα του και δεν υπάρχει απλώ η βοήθεια σε είδο η οποία ενδεχομένω να δημιουργήσει προβλήματα στην τοπική παραγωγή. Υπάρχει από ό,τι ενημερώθηκε ένα καλό παράδειγμα στον Νίγηρα και στο Τσάντ. Είναι γενικά στην φιλοσοφία του προγράμματος Αζίρ στην περιοχή Σαχέλ. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο ότι πρέπει να προσεχθεί πάση θυσία και να διασφαλιστεί η τοπική παραγωγή. Γιατί είναι ένας κύκλος. Εάν σε αυτόν τον κύκλο δεν είμαστε θετικοί και σπάσουμε μια λυσίδα θα δημιουργηθούν προβλήματα εκ των υστέρων. Φαίνεται ότι η επιλογή τουλάχιστον cash και voucher μέχρι τώρα αποδίδει. Βέβαια είναι θέμα συνθηκό. Δεν είναι πανάκια. Αλλά θα πρέπει να την λάβουμε σοβαρά υπόψη σε όλα αυτά τα προγράμματα με στόχο να εξασφαλίσουμε την τοπική παραγωγή, τους, τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς παραγωγούς. Εξάλλου είναι μέρος της ίδιας της λογικής του LRRT. Ανακούφιση, αποκατάσταση και ανάπτυξη. Αυτή η διαδικασία δεν πρέπει με τίποτα να σπάζει στη μέση. Και θεωρώ ότι το voucher και το cash μέχρι τώρα από ό,τι έχουν ενημερωθεί αποδίδει και θα πρέπει να συνεχιστεί. Thank you, Mr. for the... Ο κύριος Κοράου από την ε, Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία βασιζόμαστε συνήθως στη συνεισφορά των πολιτών των κρατών μελών για την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρουν όμως πού θα καταλήξουν αυτά τα χρήματα, πώς θα δαπανηθούν. Επίσης, μέσα στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών και των φυσικών καταστροφών υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία για να ξέρουμε πώς ε, δίνονται, πώς χορηγούνται τα χρήματα των φορολογουμένων, δηλαδή ποια είναι τα απτά αποτελέσματα. Η διαφάνεια είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς αν διοριστείτε θα αναλάβετε δράση για διαφάνεια στον ε, τομέα της αρρωγής αυτής και θα ενημερώνετε τους πολίτες για το πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. Ποια θα είναι τα απτά αποτελέσματα στα οποία ελπίζετε να φτάσετε. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάθεση των κονδυλίων. Είπα και πριν στην απάντησή μου στον κύριο Χρυσόγωνο ότι εμφανίστηκαν προβλήματα, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα σταμάτησαν και προγράμματα ακριβώς διότι υπήρχε διαφθορά και απάτη. Αλλά η ενημέρωση μου τουλάχιστον με έπεισε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου σε τρία επίπεδα είναι ικανοποιητικοί. Και σίγουρα πάντα το κάθε τι πρέπει να τη χάνει βελτίωση με νέα δεδομένα που εμφανίζονται. Αλλά φαίνεται ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν, υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάθεση των κονδυλίων και θα πρέπει να συνεχίσει. Κάποιες αξιολογήσεις που έλαβα γνώση θεωρούν τουλάχιστον ότι στο επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΧΟ υπάρχει σωστή διάθεση των κοντιλίων που φτάνει στα πιο ψηλά επίπεδα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν είμαι αφελής, επαναλαμβάνω, να πιστεύω ότι δεν θα εμφανιστούν θέματα διαφθοράς και απάτης. Δεν θέλω να πω ότι οι σημερινοί μηχανισμοί είναι τέλειοι, αλλά φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικοί. Εάν στη διάρκεια των αξιολογήσεων που γίνεται ακόμα και από ιδιωτικούς εμπειρογνώμονες προκύψει οποιαδήποτε αντίληψη και αξιολόγηση που οδηγεί σε βελτίωση της όλης διαδικασίας, σαφέστατα πρέπει να προχωρήσουμε στην βελτίωση τη διαδικασία για να μην χάνονται τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα των προπολογισμών, διότι ειδικά σε περίοδο οικονομική κρίση και είμαι από χώρα που περνά οικονομική κρίση, δεν πρέπει να, να χάνονται καθόλου λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλιό από τους μη εγγεγραμμένους. Κύριε Επίτροπε, αγαπητέ συνάδελφε, μιλάμε για πόλεμο, κρίση, πανδημία, φυσικές καταστροφές. Στην ουσία είμαστε οι πυροσβέστες ορισμένων πολιτικών ή καταστάσεων ή απορριθμίσεων, φυσικών απορριθμίσεων. Αλλά φέρουμε μεγάλη ευθύνη ως προσωρισμένα φαινόμενα ή καταστροφές, δηλαδή τους, 3.000 μετανάστες που πνίγηκαν στη Μεσόγειο και την ευθύνη της δύση. Είμαστε ουραγοί των Αμερικανών πολλές φορές και πολλές φορές υπάρχει μεγάλη διαφθορά και εμείς εφησυχάζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε καλές σχέσεις με χώρες που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο και που πληρώνουν τις συνέπειες της πολιτικής τους ή που δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις έναντι των πληθυσμών τους τους οποίους εμείς υπερασπιζόμαστε ποια μέσα διαθέτεται ως επίτροπος για να ε, ελέγξετε την αποτελεσματικότητα της δράσης μας, ιδιαίτερα στις μεγάλες κρίσεις της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Κύριε συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σε πολλά που είπατε, δεν θα έλεγα ότι είμαι σύμφωνος, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις σας. Και είπα, θα μιλώ ως πολιτικός με πολιτικούς και η ειλικρίνεια είναι η πιο καθαρή βάση της συνεργασίας και της συνεννόησης. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική δράση, που ενδιαφέρει τον Επίτροπο Ανθρωπιστικής Δράσης, θα πρέπει όντως με κάθε μέσο να διατηρήσει τις τέσσερις βασικές αρχές για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στα θύματα, να τους προσφέρει τη βοήθεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πολιτικής λειτουργίας. Ανεξαρτήτως από οποιασδήποτε ευρωπαϊκές πολιτικές υπάρχουν σε συγκεκριμένα θέματα και επιδιώκουν να λύσουν τα προβλήματα περιορίζοντας τις ρίζες των προβλημάτων. Ακριβώς γι' αυτό όρισα ως βασική φιλοσοφία τη συνέχιση της πολιτικής της κυρίας Γεωργίευα το in but out. Ναι, στα θέματα του comprehensive approach, της ολιστικής προσέγγισης, θα είμαστε in, αλλά την ίδια στιγμή, για να διαφυλάξουμε την ανθρωπιστική δράση, θα πρέπει να είμαστε και out. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αυτή η διασφάλιση της ανθρωπιστικής δράσης εξασφαλίζοντας τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας του ανθρωπισμού είναι η πρόσβαση προς τα θύματα. Συμμετέχουμε στη πολιτική, δίνουμε τα στοιχεία μας, συμμετέχουμε στο project team, όπως το όρισε ο πρόεδρος Γιούνκερ, αλλά την ίδια στιγμή διασφαλίζουμε απόλυτα τη δυνατότητα ανθρωπιστικής δράσης. Είναι αξίωμα για την ανθρωπιστική δράση. Εάν το χάσει αυτό, ουσιαστικά χάνει την ύπαρξή της. Σα um, Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ζαμπορφσκά για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τις τελευταίες ημέρες Μιλάμε για την Συρία στα πλαίσια της κρίσης των προσφύγων και για το Ιράκ. Κατά τα τρία τελευταία χρόνια είχαμε έναν πόλεμο που εξελίχθηκε σε εμφύλιο και 9 εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ. Οι τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους ε, ανάγκασαν χριστιανούς και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες να καταφύγουν και να εκτοπιστούν, να καταφύγουν αλλού και να εκτοπιστούν. Θεωρείτε ότι έχουμε επαρκή ε, μέσα σε όγκο και αποτελεσματικότητα για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες ε, της ε, Συρίας και του Ιράκ για να μπορέσουν να επιβιώσουν ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα σύραξη που θα συνεχιστεί. στην περιγραφή της κατάστασης. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό ενδεχομένω και η προκάτοχός μου, συνάδελφος κυρία Κρυσταλλίνα Γεωργίευα, έκανε ειδική επίσκεψη στο Κουρδιστάν, στο Ενμπίλ, ακριβώς για να δει επιτόπου την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά και τους πρόσφυγες, αλλά σε ό,τι αφορά και τις μειονότητες θρησκευτικέ και άλλες. Και η δράση δυστυχώς της ISIS είναι όπως την έχουμε δει όλοι και μέσα από τα social media δυστυχώς. Λοιπόν, ε, χρειάζεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα που έρχεται και ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η διαχείμαση στην περιοχή του Κουρδιστάν χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οργάνωσης αυτής της διαχείμασης. Οργάνωση των προσφύγων και είμαστε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, σε συνεργασία με, τους, με τα UN agencies, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα για να εξασφαλιστεί η ζωή αυτών των ανθρώπων, των παιδιών τους και των ευάλωτων άλλων ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη γι' αυτό τον λόγο έχει δημιουργήσει γραφείο στο ΕΛΜΠΙΛ για να είναι κοντά. Να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση και να την καταγράφει έτσι ώστε να έχει την πιο καλή εκτίμηση δεδομένων. Έχει κινηθεί ακόμη στην περιοχή μέχρι και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για να βοηθήσει. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το αλλά τουλάχιστον περιορίζουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω συντονισμός συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους έτσι ώστε να εξασφαλιστούν και οι εθνικέ και θρησκευτικέ μειονότητε, αλλά ταυτόχρονα και οι ανάγκε των ανθρώπων εν ώψη χειμώνα στην περιοχή αυτή. Σα Σας ευχαριστώ, ο κύριος Φοντζούλικ, από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, Στυλιανίδη, όπως αναφέρατε κατά πάσα πιθανότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη της δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην διαχείριση κρίσεων. Ιδιαίτερος και ακόμα περισσότερο μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Η αναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κάτι το ξεχωριστό πλέον. Η ανθρωπιστική συνεργασία και η συνεργασία για την ανάπτυξη έχουν διαφορετικούς σκοπούς, διαφορετικές αρχές και διαφορετικές, ε, διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής. Αλλά μετά από την ανταπόκριση σε καταστάσεις ε, κατεπίγουσας ανάγκης, η κατάσταση συχνά προαπαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη για την ανάπτυξη. Πώς μπορεί λοιπόν ο συντονισμός της μετάβασης από την ανθρωπιστική βοήθεια στην μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη να βοηθήσει σύμφωνα με τη σύνδεση αρρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης και των σχετικών αρχών που αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνένεση του 2007 για την Ευρωπαϊκή αρρωγή. Πώς εσείς ως Επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και την διαχείριση κρίσεων θα συνεργαστείτε με τον Επίτροπο για την Ανάπτυξη και την είπα το εκπρόσωπο για να συντονιστούν οι πολιτικές, για να μην υπάρχουν χάσματα στην αρρωγή σε αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία. Ευχαριστώ. Αγαπητέ θέσατε ένα βασικό ζήτημα που όντως συνδέει τους δύο βασικούς άξονες του resilience building. Δηλαδή την αλληλοσυμπληρωματικότητα μεταξύ της ανθρωπιστικής δράσης και της ανάπτυξης. Ουσιαστικά ορίσατε το πλαίσιο της συνεργασίας του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Δράσης και του Επιτρόπου Ανάπτυξης. Που αυτό βασίζεται σε αυτό που είπατε τη σύνδεση του linking LRRD, τη σύνδεση της ανακούφισης, αποκατάστασης με ανάπτυξη. Εάν δεν υπάρξει ανθρωπιστική δράση η οποία θα προετοιμάσει την ανάπτυξη, θα υπάρξει πρόβλημα. Θα συνεργαστούμε με τον συνάδελφο κύριο Μίμητσα πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Και ήδη είπα ότι υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολύ γόνιμης συνεργασίας. Θα επαναλάβω το Αζίρ στο Σαχέλ, το share στη ογκέρα της Αφρικής που είναι παραδείγματα αυτής της δράσης και αυτής της αποτελεσματικότητας. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθούμε αξιολογώντας συνεχώς αυτή τη δράση. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνεχώς το accountability ως εργαλείο το οποίο θα μπορεί να μας προσφέρει ακριβώς τη, την, βελτίωση των πρακτικών. Πιστεύω ότι διατηρώντας αυτό τον κύκλο, ξεκινώντας από το εκτίμηση κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου, αντιμετώπιση και μετά εξελίσσοντας στο resilient building, μπορούμε ακριβώς πολύ σωστά να βελτιωθούμε και να κάνουμε και οικονομίες κλίμακους. Επιμένω ότι θα είμαι σε αυτή τη γραμμή, μάλιστα στη λογική ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Δίνουν τα λεφτά στην πρόληψη, κερδίζεις. Είναι ένα ευρώ στην πρόληψη, αποφεύγεις 7 ευρώ στη θεραπεία. Ο συνδυασμός δηλαδή, είναι ένα προς 7. Είναι τόσο μεγάλη η οικονομία κλίμακος. E ευχαριστώ κύριε Κάρσκι από τους Ευρωπαίους Συντελετικούς Συντακτημιστές, το ECR. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, κύριε Σιλιανίδη. Έχετε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ανθρωπιστρατιωτική δράση για να διασφαλίσετε την προστασία και την διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, οι διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις ε, χρησιμοποιούν ε, τις ε, υπηρεσίες στρατιωτικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων. Γιατί ο τρόπος δράσης τους σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να συγκριθεί με τις διεθνείς ε, επαγγελματικές οργανώσεις στρατιωτών. Ερωτώ λοιπόν, θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις επαγγελματίες στρατιώτες. Θα σας κάνω μια διευκρίνηση γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και οι εμπειρίες μέχρι τώρα μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Βασική αρχή είναι ότι ναι, αποφεύγεται η στρατιωτική δράση για ανθρωπιστική βοήθεια και αρρωγή γιατί χάνουμε την ανεξαρτησία μας, την αμεροληψία και ουδετερότητα την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε για να έχουμε άξες στα θύματα. Όμως υπήρξαν ένα-δύο παραδείγματα που η ανθρωπιστική, η στρατιωτική βοήθεια ήταν σωστική στην ανθρωπιστική δράση. Στη Λιβύη παραδείγματος χάρη όπου υπήρξε βοήθεια στρατιωτική για να σωθούν ζωές. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί διότι ακριβώς σώζουμε ζωές. Κάτι ανάλογο έγινε και στη Σομαλία. Υπάρχει όμως ένα κακό παράδειγμα. Στο Αφγανιστάν υπήρξε ανάμειξη στρατιωτικής και ανθρωπιστικής δράσης όπου δημιούργησε προβλήματα στη δυνατότητα της ανθρωπιστικής δράσης να έχει άξεις. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αυτό κρίνεται εκ των συνθήκων και των πραγμάτων. Και εδώ είναι αυτό που είπα. Ότι είμαστε πολιτικοί. Έχουμε τις αρχές, τις αξίες, αλλά έρχονται και δύσκολα διλήμματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Και εκεί θα είναι όντως ο ρόλος του Επιτρόπου. Να βρει τη λύση εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία της ανθρωπιστικής δράσης αλλά εάν προκύψει θέμα όπως τη Λιβύη που σώζει ζωές, τότε μπορεί να αξιοποιήσεις με βάση τις αρχές του Όσλο την έσχατη λύση. Μόνο τότε. Σας ευχαριστώ, η κυρία Πακαδοντούντουα από την Αλντε. Ε, ευχαριστώ και να καλωσορίσω τον κύριο Στυλιανίδη. Καταρχήν, ε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το προσωπικό σας αποτύπωμα και ελπίζω αυτό να δώσει μία όθηση στη μελλοντική σας δραστηριότητα. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι το οποίο να ε, απασχόλησε και στην ε, παρέμβαση του κυρίου Μίμητσα. το 2013 δυστυχώς πέθαναν πολλοί εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι παράγοντες ε, κινδύνου για τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια και αυτούς που εργάζονται επί επιτοπίες. Ο κύριος Μίμητσα μας είπε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα και θεωρεί ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ε, κρίσεις αυτές. Θα ήθελα να μας πείτε πώς θα έχει η διαχείριση της ασφάλειας των εργαζομένων έτσι ώστε να εγγυηθούμε τη φυσική ε, ακαιρεότητα των ε, συνεργατών αυτών που εργάζονται επιτοπίως για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε στο θέμα. Έχω ανάλογη ευαισθησία, γι' αυτό και στην αρχική μου ομιλία τίμησα τον Βρετανό ανθρωπιστή εργάτη. Όμως θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω ενημερωθεί για αυτά τα security clearance, για την κατάρτιση που γίνεται στους ανθρωπιστές, στους εργάτες αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από τα NGOs αλλά δεν έχω ειδική ενημέρωση σε ό,τι αφορά άλλα θέματα ασφάλειας αυτών των ανθρώπων. Θα ήταν εκ μέρους μου αυτή τη στιγμή προχειρότητα και θα ήταν άσοφο εάν ερασιτεχνικά μιλούσα για κάτι που δεν ξέρω καλά. Πιστεύω ότι θα ήταν λάθος. Αλλά, όπως και ο κύριος Μίμητσα, θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να καταφύγουμε στις υπηρεσίες που ξέρουν το θέμα, ενδεχομένω να χρειαστούμε και ειδική τεχνογνωσία ειδικών ανθρώπων σε αυτά τα θέματα και ο συνάδελφο πριν μίλησε για ανάλογα θέματα παραστρατηγικών οργανώσεων, πώ του αντιμετωπίζει, για να μειώσουμε τον κίνδυνο των ανθρώπων αυτό. Υπάρχει κάτι σε εξέλιξη που θέλω να το πω και με ενθαρρύνει. Υπάρχει εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία την εθελοντική. Φαίνεται ότι εκεί μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εάν αυτοί οι εθελοντέ μα οι οποίοι ελπίζω να είναι πολύ σύντομα στην εφαρμογή του προγράμματος και να συμμετάσχουν στην όλη ανθρωπιστική δράση. Εξειδικευτούν κάποιοι από αυτούς τα, αυτά τα θέματα, ίσως να βοηθήσουν πολύ τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε αυτόν τον τομέα. Λέω ιδέες τώρα που ε, εμφανίζονται εξαιτία όλων αυτών που έχω ενημερωθεί. Σας λέω πρέπει να γίνει πολύ πιο συστηματική δουλειά ακριβώς σε αυτά τα θέματα της ασφάλειας. Ε, Κύριε Χρυσόγονος, πριν από πίσω σα Κύριε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θαραλέα πραγματικά υπόσχεσή σας ότι εφόσον επιβεβαιωθείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταβείτε αυτοπροσώπως στις χώρες της Αφρικής που πλήττονται από τον ιό έμπολα για να εκτιμήσετε επιτόπου την κατάσταση. Διότι πιστεύω ότι ο Επίτροπος προκειμένου να επιτελέσει τον επιτελικό του ρόλο θα πρέπει κάποιες στιγμές να βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών καταστροφών ή αναγκών. Μπορείτε να μας βεβαιώσετε από τώρα ότι η δέσμευσή σας για αυτοπρόσωπη μετάβαση ισχύει εξίσου και για κάθε άλλη περίπτωση σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που μπορεί να ανακύψει κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Κύριε συνάδελφε, όπως λέμε και στα ελληνικά, εγώ δεν, λέω κουβέντες του αέρα. Όταν λέω κάτι το εννοώ. Και η δέσμευση είναι δέσμευση. Και έτσι πρέπει να είναι η πολιτική δέσμευση μπροστά σε μια τέτοια επιτροπή. Προς Θεού να λέμε κάτι που δεν θα κάνουμε. Μετά χάνουμε πλήρως την όποια αξιοπιστία έχουμε ως πολιτική. Γι' αυτό, ναι, το πρώτο ταξίδι θα πρέπει να είναι στις περιοχές του έμπολα που πλήττονται. Ακριβώς για να δω επιτέπου τι γίνεται, αλλά και να σταλεί συμβολικό μήνυμα. Και σας λέω, στο θέμα της παρουσίας περισσότερου ιατρικού προσωπικού, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αυτό το συμβολικό, μήνυμα. Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί έχουν στήσει κάποια νοσοκομεία και έχουν έρθει και σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου για να υπάρξει και από πλευρά Κυπρίων γιατρών τέτοια ενίσχυση. Το θεωρώ προσωπική μου συμβολή. Όντα ω Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για Ανθρωπιστική Δράση, όταν θα είμαι εκεί, στέλνω το μήνυμα στου συναδέλφου μου γιατρού τη Κύπρου ότι πρέπει να πάνε να βοηθήσουν σε αυτό το νοσοκομείο. Λέω κάτι που το νιώθω ω ένα απλό παράδειγμα γύρω από αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό, εκτό από την πρακτική αξία που θα μπορέσω να συντονίσω, να καταγράψω άμεσε ανάγκε και να μπορέσω όντω να κινητοποιήσω πράγματα, επιμένω και σε αυτή τη συμβολική σημασία ότι ναι, οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται από τη στιγμή βέβαια που θα έχουν τη δυνατότητα του evacuation. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γράψατε στην επιστολή σα ότι ναι, όλα αυτά έχουν μια προπόθεση. Το evacuation. Αλλιώ είναι άδικο να πάρουμε κόσμο στο λαιμό μα. Είναι άδικο να στείλουμε κόσμο εάν δεν τον εξασφαλίσουμε σε επίπεδο μάλιστα ιατρικού προσωπικού. Thank um, ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Σαρτζεντίνη από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Μιλήσατε για τις ξεχασμένες κρίσεις. Θα ήθελα να μιλήσω για ξεχασμένους λαούς, λαούς που έχουν μείνει πίσω. Λαοί που μπορούμε να δούμε, στους οποίους δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Στο Γιαρμούκ, στη Συρία για παράδειγμα, για Σίντι, το ε, όρο Σινιάν. Υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε καν, Λαοί που δεν μπορούμε να τα δούμε στο κράτος του Πλενήλου, στο Νούμπα, στους Νούμπα στο Σουδάν. Ύστερα υπάρχουν λαοί, άτομα τα οποία μπορούμε να έχουμε, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, αλλά δεν μπορούμε να τους δούμε. Για παράδειγμα, άτομα τα οποία ζουν σε περιοχές όπου δεν φτάνει η αρρωγή, το Ανατολικό Κονγκό στο κόμμα ε, στο Βόρειο Κιμπού, κοντά στο Γκόμα υπάρχει διεθνής ε, αρρωγή και υποστήριξη, αλλά λίγο πιο πάνω δεν υπάρχει κανείς. Και υπάρχουν άτομα στα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι κυβερνήσεις, οι αντάρτες και άτομα στα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε γιατί πολύ απλά δεν καταβάλουμε προσπάθεια να πάμε παρακάτω. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι ο ανθρωπιστικός χώρος συρρυκνώνεται. Άρα ερωτώ συνολικά τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την τάση του συρρυκνόμενου χώρου της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της, του περιορισμού του ανθρωπιστικού χώρου. Το πρόβλημα της πρόσβασης στα θύματα, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όντως είναι ένα θέμα που δεν έχει εύκολη λύση για να είμαστε ειλικρινεί. Είναι εδώ που λέμε ότι στα ανθρωπιστικά προβλήματα πρέπει να έχουμε πολιτικές λύσεις για να μπορέσουμε όντως να φτάσουμε στην καρδιά του προβλήματος. Όμως θα έλεγα ακριβώς εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας βασική μου αρχή για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα θύματα θα είναι ότι θα είμαι έτοιμος να συνομιλήσω ακόμα και με τον διάβολο. Ναι, πρέπει να βρούμε τρόπο να διαβουλευτούμε για να πάμε. Αλλιώς θα μιλούμε θεωρητικά. Και πιστεύω ότι ναι, πρέπει ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δράσης να είναι έτοιμος να κάνει τέτοιου είδους συνομιλίες. Γι' αυτό πρέπει να κρατεί την αξιοπιστία του στο επίπεδο των αρχών της ανθρωπιστικής δράσης να συνομιλήσει και με τον διάβολο για να μπορέσει ακριβώς είτε να τον πείσει είτε να του επιβάλλει εκ των πραγμάτων την πρόσβαση στα θύματα που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Thank you. Ε, σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκίλ από το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε για την πειρατεία στο κέρας της Αφρικής που προκαλείται από την υπεραλίευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σπρώχνει τους Σομαλούς στην πειρατεία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ευρέα δεδομένο, δεδομένο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπήρξε αύξηση 42% στις επιθέσεις πειρατείας στον κόλπο της Γουινέας και οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι οι πειρατείες είναι πολύ πιο βίαιοι γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ουσιαστικά να ληστεύσουν και όχι τα λίτρα. Πολλοί από τους πειρατές αυτούς λοιπόν είναι πρώην αλληλείς, ψαράδες που έχουν δει το βιός να, καρα... καταστρέφεται από την υπεραλίευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί σοκ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει το ρόλο που έπαιξε στερώντας τους πόρους αυτούς από, το... την Αφρική. Σε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού... που παρουσιάστηκε στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται ότι είναι ανησυχητικό το ποια πολιτική ακολουθείται στην, στην Αφρική σε ό,τι αφορά την Αφρική, στο κέρας της Αφρικής. Και τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε τίποτα και τώρα υπάρχει απειλή αυτή. Στην ε, ε επιστολή του κ. Γιάνκουν αναφέρεται ότι οι προτεραιότητες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τροποποιηθούν, να μεταρρυθμιστούν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μετά από έξι έτη προειδοποιήσεων η πρώην Επίτροπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έκανε τίποτα και ίσως να σχολιάσετε και την δική σας στρατηγική. Αγαπητέ συνάδελφε είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα και οι λεπτομέρειες που αναφέρετε είναι εκτός της ενημέρωσής μου για να είμαι ειλικρινή. Είναι ένα θέμα που δεν έχω ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τα θέματα υπεραλίευση και δεν εμπίπτουν και στα πλαίσια του, του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου ανθρωπιστική δράση. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή τη Σομαλίας, παρόλα τα πολύ σημαντικά πολιτικά προβλήματα που υπάρχουν και υπάρχουν φοβεροί κίνδυνοι δυστυχώς από, την, από τον υποσυντισμό, από την έλλειψη βασικών αναγκών. Υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι που έχει παραχωρηθεί στην περιοχή ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους πληθυσμούς που έχουν αυτή την ανάγκη. Είπα και πριν και δύο-τρεις φορές το πρόγραμμα SHARE που ασχολείται ακριβώς συνολικά με το κέρας της Αφρικής και τη Σομαλία για να βάλει την όλη περιοχή μέσα σε μια λογική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να υποτιμείται, να υποτιμηθεί ως ευρωπαϊκή πολιτική για να μπορέσουν οι πληθυσμοί εκεί να μπουν σε μια διαδικασία αποκατάστασης ανάπτυξης. Τώρα, κάποια θέματα που αναφέρετε, οφείλω να μου ότι δεν ξέρουν θέματα υπεραλίευσης, δεν έχω ενημερωθεί για αυτά. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλά στην περιοχή ως βασικός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας και θα έλεγα ότι ε, πρέπει να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα. Τώρα, μέσα στα περιορισμένα βέβαια πλαίσια ενός προϋπολογισμού. Τώρα, τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα με τα οποία δεν μπορώ να σχοληθώ να συζητήσω και θα ήταν λάθος να μπω σε θέματα που δεν ξέρω πολύ καλά τις λεπτομέρειες τους. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Γιάνσεν από τους μη εγγυγραμμένους. Πρόεδρε, η επιστημιστική αρρωγή είναι κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο. Η επιστημιστική αρρωγή σε κάποιες περιπτώσεις όμως αφαιρεί το βιός ε, των τελευταίων ε, παραγωγών τροφίμων επιτόπου. Με άλλα λόγια, αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως. Και συνέπεια αυτού είναι πραγματικά μια επιστηστική κρίση η οποία συνεχίζεται επί χρόνια και χρόνια. Γιατί έχει χαλάσει η αλυσίδα μέσω της αρρωγής ε, της ανθρωπιστικής. Μπορεί ο υποψήφιος να μας εγγυηθεί ή να υποπτεύσει σε περίπτωση που χρειαστεί να παρασχεθεί κάπου επιστηστική αρρωγή, δεν θα καταστραφεί η δυνατότητα παραγωγής των τελευταίων τοπικών παραγωγών. Έχω ήδη αναφέρει το παράδειγμα του Αζίρ ως προγράμματος του Σάχελ. Ακριβώς που είχε αυτή την ειδική ευαισθησία το όλο πρόγραμμα να λάβει υπόψη του κατά κύριο λόγο την τοπική παραγωγή. Και έχω πει και την εξέλιξη στην επιστημιστική βοήθεια που βασίζεται στη φιλοσοφία των vouchers και του cash. Ακριβώς για να δώσει τη δυνατότητα ο άνθρωπος που δέχεται τη βοήθεια να παίρνει τοπικά προϊόντα, να αγοράζει τοπικά προϊόντα. Να μην χρειάζεται δηλαδή να είμαστε στην παραδοσιακή μέθοδο όπου δίνεται βοήθεια σε είδο και πολλές φορές δεν έφτανε και στον άνθρωπο που την είχε ανάγκη. Και μετά από αξιολογήσεις από ό,τι με έχει ενημερώσει η ΕΚΟ υπήρχαν όντως πολλά προβλήματα. Δεν λέω ότι είναι πανάκια επαναλαμβάνω. Είναι θέμα συνθήκο. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας του resilience building αυτό το θέμα που αναφέρεται είναι βασική πρωταρχική αρχή. Ότι ναι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έτσι ώστε η βοήθεια που προσφέρεται να μην επηρεάζει σε καμία περίπτωση την τοπική παραγωγή. Είναι θέμα που πιστεύω ότι το σέβεται η λογική της ανθεκτικότητας του ρεζίλιας και είναι ακριβώς η μια καινοτόμα φιλοσοφία γύρω από την βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα έλεγα θα πρέπει στους ανθρώπους που σκέφτηκαν όλες αυτές τις καινοτόμες ιδέες και τα προγράμματα να τους πιστώσουμε με μια πολύ σοβαρή εμπειρία και τεχνογνωσία. Γιατί είναι χρόνια που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Και με ένα τουλάχιστον με έχει πείσει η όλη μου ενημέρωση γύρω από αυτά τα θέματα του resilience building ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να συνεχίσει και αν είναι δυνατόν να επεκτηθεί και να δοθεί πάλι στα περισσότερο βάρος στον προϋπολογισμό των όλων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Σας ευχαριστώ κύριος Χέι από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον υποψήφιο Επίτροπο στην Ακρόαση να τον ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που μας έχει δώσει στις ερωτήσεις μας. Όπως καλά θα γνωρίζει, η αντιμετώπιση των κρίσεων αποτελεί ένα θέμα που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις ερωτήσεις έχω για σας. Καταρχάς, η Ευρώπη είναι πλούσια και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ως Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν τόσο εκπληκτική εργασία ανθρωπιστικής φύσεως. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη δέσμευση με τον κλάδο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική αρρωγή. Κατά δεύτερον, υπάρχει μεταρρύθμιση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου του 2016. Ποια θέματα θα θέσετε επιτάπητο για να μεταρρυθμίσουμε το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα άνωτα όρια για την ανθρωπιστική αρρωγή. Γιατί ένα χρόνο έχουμε ακόμα. Και τρίτον, θα δεσμευτείτε σε ό,τι αφορά την προβλεψιμότητα και την ε, έγκαιρη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής αρρωγής προκειμένου ως Επίτροπος να δώσετε την ε, βεβαίωση αυτή προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις άλλες οργανώσεις που δεσμεύονται για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε συνάδελφε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το βασικό είναι να καταφέρουμε την εξισορρόπηση payment and commitments. Είναι βασική θέση και αρχή. Γι' αυτό είναι πρώτη στο στόχος. Πρέπει και στα πλαίσια του κολεγίου, ως Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δράσης, με τη δική σας βοήθεια, και τη χρειαζόμαστε, σας λέω ειλικρινά, να πείσουμε για την ιδιαιτερότητα της ανθρωπιστικής δράσης. Και να μπορούμε, όπως σωστά είπετε, να χρηματοδοτούμε τις εξαιρετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις τις δικές μας ευρωπαϊκές για να συνεργάζονται με τοπικές στην Αφρική, στην Ασία, οπουδήποτε, στη Συρία, στο Ιράκ για να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει αυτό να είναι επιδίωξη, θα έλεγα και πριν από το αναθεώρηση του MFF το 2016. Είναι στόχος συνεχόμενος. Είναι στόχος που τίθεται από τώρα. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή απόφαση τη σημερινή έγκριση από την Budget Committee γύρω από το θέμα αυτό. Ήδη το Κοινοβούλιο στηρίζει αυτό το πράγμα. Είναι μια, ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να πάρουμε. Είχατε κάνει ενέργεια ως, ως Είχε σταλεί επιστολή από τις 10 Σεπτεμβρίου ακριβώς για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της εξισορρόπησης των payments και των commitments. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια που είναι κοινή και εσείς και εγώ αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξισορροπήσουμε το συντομότερο τα payments με τα commitments για να μπορούμε να αποδίδουμε στι μη κυβερνητικέ οργανώσει όσα χρειάζονται και να μπορούν να δρουν. Αλλιώ δεν θα μπορούν να δρουν. Για να διατηρήσουμε τον κύριο μα παγκοσμίω, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε και οι διεθνεί μα εταίροι, τα UN agencies, να μα έχουν εμπιστοσύνη. Συμφωνώ πολύ Thank you. And our next question is... Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Σλάιν από τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Οι καταστροφές είναι φυσικές καταστροφές πολλές φορές που δεν μπορούν να αποφευχθούν. Θα μπορούσαν όμως να αποφευχθούν με την ε, πρόληψη. Το 2013 το 20% των δραστηριοτήτων της ΕΚΟ ε, αφορούσαν την πρόληψη γιατί έτσι μπορούμε να σώσουμε ζωές, να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα και το κόστος μπορεί να είναι αποδοτικό. Για να ε, μειώσουμε λοιπόν για να μειώσουμε τις καταστροφές θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θέση μας και στην διάσκεψη που θα γίνει του χρόνου στην Ιαπωνία. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να δράσουμε σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο μέσα στα πλαίσια της πρόληψης. Πολύ σωστά κυρία συνάδελφε είπατε ναι ότι το 2013 το 20% του προϋπολογισμού της ΕΚΟ πήγαινε στην πρόληψη και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε και πριν ότι ένα ευρώ για την πρόληψη γλιτώνει 7 ευρώ από την αντιμετώπιση της καταστροφής. Είναι η οικονομία κλίμακος εκτός των άλλων και μας δίνει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αλλού τα λεφτά. Αυτό σε κάποιο βαθμό πρέπει να το έχουμε ως πηξίδα. Και θέσατε πολύ σωστά και την επόμενη διάσκεψη του Σεντάι το Μάρτι του 2015 που θα συζητηθεί η το Hyogo Framework Action. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή θέση. Αυτή η ευρωπαϊκή θέση πρέπει να είναι θέση και του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Δράσης και της Επιτροπής. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε συνεχή διαβούλευση. Πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για να φτάσουμε σε αυτή την κοινή θέση την ευρωπαϊκή που θα είναι και πολύ έντονη θέση. Γιατί θα, θα έχει το βάρος και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ε, να βρούμε τη διαδικασία, workshop, είπα κάποιες ιδέες πριν, αυτά είναι θέματα διαδικαστικά, θα τα συζητήσουμε για να βρούμε αυτή τη λύση, να πάμε στο Σεντάι, να πάει ο Επίτροπος στο Σεντάι και να έχει την κοινή ευρωπαϊκή θέση με τη στήριξη της Επιτροπής έτσι ώστε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή του resilience building και της πρόληψης. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Είδα ικανότατο προσωπικό στην ΕΚΟ που κινείται σε αυτή τη γραμμή. Πιστεύω ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και μπορούμε ακριβώς μέσα στα πλαίσια των μεγάλων δυσκολιών των νέων ανθρωπιστικών κρίσεων τουλάχιστον να κάνουμε ό,τι μπορούμε δυνατό για να νιώθουμε κι εμείς ήσυχοι με τη συνείδησή μας. Ευχαριστώ κύριε Λούκε από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση ακόμα για, τον... Ε, τα φάρμακα σε καταστάσεις εκτάκτης, έκτακτης κρίσης. Ε, σε καταστάσεις όπου υπάρχουν ε, επιδημίες ενδεχόμενο και κίνδυνος ε, επιδημιών. Υπάρχει ανάγκη χρήσης αντιβιωτικών, αλλά ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αντιβιωτικά δεν δρούν πλέον γιατί έχουν ε, χάσει, υπάρχει ανθεκτικότητα. Και επίσης υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα επιτόπου που βοηθούν τον άνθρωπο. Ποια μέτρα λοιπόν μπορεί στον τομέα της αρμοδιότητάς σας να πάρετε, προκειμένου προληπτικά εγκαίρως να φροντίσετε όπου υπάρχουν τέτοιες ανθεκτικότητες για να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά φάρμακα. Και κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη τέτοιων φαρμάκων. Γιατί νομίζω ότι 15 έως 20 χρόνια χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου διδυτικού. με έχετε επαναφέρει στα πανεπιστημιακά μου χρόνια. όπου γινόταν συζήτηση για την εναλλακτική ιατρική και την κλασική ιατρική με τα παραδοσιακά φάρμακα. Σαφέστατα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μιλήσουμε και με τον Επίτροπο Υγείας που θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχω ήδη κάνει μια συζήτηση, συνάντηση μαζί του και στο θέμα του έμπολα και ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και επικοδομητική γιατί είναι γιατρός. Όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα μικρόβια από τα παραδοσιακά αντιβιωτικά. Και το ξέρουμε όλοι. Πιστεύω όμως ότι οι εξειδικευμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με το θέμα στις περιπτώσεις αξιολόγησης ενός μικροβίου ή ενός ιού θα πρέπει να γίνονται οι διάφορες χημικές και άλλες αναλύσεις έτσι ώστε να δίνεται ένα αντιβιωτικό που μπορεί όντως να δράσει και να είναι αποτελεσματικό. Τα θέματα εναλλακτική φαρμακολογίας είναι ένα θέμα που έχει σχέση με τον τοπικό παράγοντα. Σίγουρα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τον τοπικό παράγοντα δεν πρέπει να αποκλειστεί ή οποιαδήποτε εναλλακτική ιατρική μέθοδος. Και ξέρω ότι στην Αφρική τέτοιες μέθοδοι εξαιτίας και της κοινωνικής πεποίθησης του πληθυσμού πολλές φορές έχουν σημασία στην θεραπεία λόγω, της λόγω του ψυχολογικού υποβάθρου. Δεν θα περίπτα μια τέτοια... Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι περισσότερο θέμα να γίνει μια σωστή ανάλυση όλων των δεδομένων με βάση ιατρικά δεδομένα και είναι θέμα εξειδίκευσης μη κυβερνητικών οργανώσεων. Thank you. Our next speaker... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Γκέρενς από τους ε, Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε υποψήφι Επίτροπε, είπατε πολλές φορές ότι το πρώτο σας ταξίδι, η πρώτη σας επίσκεψη θα σας οδηγεί σε μια χώρα που έχει πληγεί από το, από το έμπολα. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Το Νοέμβριο θα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός των θυμάτων. Η κρίση άρχισε το Μάρτιο και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας άργησε και δεν ήταν στο ύψος της πρόκλησης. Δεν νομίζετε ότι χρειάζεται μία αποτίμηση της ε, λειτουργίας του ε, πολυμερού συστήματος υγείας, διότι υπάρχει μεγάλος φόρτος και βραδύτητα στην αντιμετώπιση. Δεν πιστεύετε ότι το δεύτερό σας ταξίδι θα πρέπει να γίνει στη Γενέβη για να μιλήσετε όπως πρέπει με θάρρος στη διεθνή κοινότητα. Εγώ είμαι φανατικός του συστήματος, του πολυμερού συστήματος, αλλά θα πρέπει να μπει τάξη. Η κρίση μας οδηγεί σε ε, λογοδοσία και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό δεν θα πρέπει να αναφέρεται στη Γενέβη. Έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από τον πρόεδρο Ομπάμα και ουσιαστικά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας παραδέχεται αυτή την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του έμπολα. Θα ήθελα όμως για να είμαι δίκαιος να πω ότι η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα από τον Μάρτιο είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου στέλνοντας τα πρώτα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή έστειλε το μήνυμα πρώτη και πρέπει να το πούμε για να είμαστε δίκοι στην ανάλυση και στη λογοδοσία που πολύ σωστά αναφέρεται. Και έχετε δίκιο, ναι, ότι πρέπει σε επίπεδο διεθνού συστήματο πολυμερού και τα θέματα υγεία πρέπει να υποθούν τα πράγματα με ένα καθαρό τρόπο. Γιατί αργήσαμε. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Βάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ναι, το πρώτο ταξίδι θα πρέπει να είναι στις πληγήσεις περιοχές, ακριβώς γιατί σημασία έχει τώρα όχι τόσο η λογοδοσία, όσο το τι κάνουμε στην πράξη. Σημασία έχει να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει, διότι είναι έξω από τα σπίτια μας, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και όπως είπε, είπα και πριν ο επιδημιολόγος, πρόεδρος της World Bank, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια μορφή επιδημία. Γι' αυτό πιστεύω ότι ναι, η επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές θα βοηθήσει στην συνέχιση της κινητοποίησης, της εγρήγορσης και στην πρακτική συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατροί επιτόπου, νοσηλευτικό προσωπικό επιτόπου, κλινικές κινητές μονάδες, θεραπεία και σιγά σιγά αποκατάσταση των συστημάτων υγείας των συγκεκριμένων χωρών. Διότι εάν δεν γίνει αυτή η αποκατάσταση ταυτόχρονα, ουσιαστικά θα χτίζουμε στην άμμο. Χρειάζεται να κινούμαστε και με την αποκατάσταση των συστημάτων υγείας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να επενθυμίσω ότι πρέπει να τηρούμε το χρονικό διάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, γιατί έχουμε αργήσει 10 λεπτά. Η κυρία Σάντσες Κάλεν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή είσαστε Κύπριος και έχετε μία ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα, όπως ξέρετε το 11-12 η Παλαιστίνη έλαβε 275 εκατομμύρια ε, ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 15 νοσοκομεία χρειάστηκε να κλείσουν και 25 σχολεία καταστράφηκαν. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποδοθεί ευθύνη στους Ισραηλινούς αυτή την ε, ε, σύραξη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να χτιστούν αυτά τα νοσοκομεία και τα σχολεία δόθηκε βοήθεια και χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Δεν θα πρέπει λοιπόν η ανθρωπιστική βοήθεια να δίδεται άμεσα στους Παλαιστινίους χωρίς να μεσολαβεί το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά σε αυτές τις περιοχές των μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων τώρα, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, οι χώρες γύρω από την περιοχή υφίστανται πολύ μεγάλο κόστος. Η Τουρκία, είπα πριν, ο Λίβανος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου το κράτος δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει να αντέχει αυτό το μεγάλο όγκο προσφύγων μιλάμε για ένα γεωπολιτικό σοκ. Γι' αυτό πρέπει πάση θυσία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Απλώς ως παρένθεση για αυτό που αναφέρεται για την κυπριακή μου καταγωγή. Επί της ουσίας, είναι γεγονός ότι στην περιοχή C, στην περιοχή Γ, οι κοδομές που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταστραφεί. Και Ήδη όπως γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτησε αποζημίωση από το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι σωστό. Και πρέπει αυτή η απέτηση να συνεχίσει. Δεν μπορεί τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων που δίνονται για αποκατάσταση ανθρωπιστικής βοήθειας να υφίστανται αυτή τη μεταχείριση. σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής, αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε επίτροπος θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα με βάση τις βαθύτερες αιτίες. Η απόφαση της, 30, Αυγούστου, πριν ένα μήνα ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά την εκεχηρία στη Γάζα, ήταν καθαρή και σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα δύο κράτη, Ισραήλ και Παλαιστίνη, στηρίζει την εγκεχηρία και ελπίζουμε να συνεχίσει και να έχει πρόσβαση. Συγχωρείτε, τελείωσε ο χρόνο. Θα έχετε χρόνο στο τέλο, σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει κάτι. Η κυρία Χάιμπουχ για του πράσινου. Καταρχά, κυρία Στυλιανίδη θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ βάθου καρδία για τη συνδέσμευσή σα. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μια κοινή θεώρηση και αυτό είναι βασική προπόθεση. Αλλά παρά τι προσπάθειες που έγιναν σε όλα τα επίπεδα, πάντα υπάρχει η κριτική για τη συνεργασία με τις τοπικέ δομέ στα πλαίσια τη ανθρωπιστική βοήθεια. Ότι αυτό είναι κάτι το οποίο παραμελούμε και δεν το προωθούμε ενεργά. Πώς λοιπόν προτίθεστε αυτή την αποτυχία της ανθρωπιστικής βοήθειας να την βελτιώσετε στο μέλλον. Τι προτίθεστε να κάνετε για την μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο μέλλον. Θέλω να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης για αυτό το θέμα της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες με βάση την ενημέρωσή μου για να μπορέσουμε έτσι να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο καθαρά. Η ενημέρωση μου λέει ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι ευρωπαϊκέ, έχουν επαφή και συνεργασία με τοπικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα διότι υπάρχει θέμα κριτηρίων σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο know-how και εκεί είναι το πρόβλημα της απευθείας ουσιαστικά επαφής. Και υπάρχει και νομοθεσία βέβαια που επιβάλλει τη συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά είναι το πλαίσιο και τα πρακτικά ζητήματα. Τώρα, η πληροφόρηση μου εμένα τουλάχιστον μου λέει ότι ναι, υπάρχει απόλυτη συνεργασία και ίσα ίσα μόνο εάν υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες τους local actors μπορεί και αποδίδει η δουλειά των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω εσείς υπονοείτε ότι δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα το κοιτάξω σε συγκεκριμένη βάση, σε ποια περιοχή, πού, για να διερευνήσω εάν αυτό το θέμα έχει σχέση με τοπικές συνθήκες και δεν είναι γενικό πρόβλημα. Γιατί εάν αποδεχτούμε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε περνούν από τόσα κριτήρια αξιολόγηση, δεν έχουν διάθεση να συνεργαστούν με τοπικού παράγοντε, σημαίνει κάπου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά αν είναι σε τοπικό επίπεδο, σε συγκεκριμένη περιοχή, χώρα, τότε ναι, πρέπει να δούμε τη λύση επιτόπου. Ομολογώ ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε επιτόπου και εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας θα είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και να μου υποδείξετε για να πάω να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη από την Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Είναι παρούσα Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ε, σειράξεις που σχετίζονται και που οδηγούν μάλλον και σε περιβαλλοντικές ε, καταστροφές ή κλιματικές ε, αλλαγές θα δημιουργήσουν προβλήματα στους υδάτινους πόρους που είναι χρόνιο πρόβλημα για αυτές τις χώρες. Το 2007-12 για στον τομέα αυτό έπρεπε να χορηγήσουμε 2 δις 200 εκατομμύρια ευρώ για να προσπορήσουμε υδάτινους σπόρους και να αντιμετωπίσουμε την κρίση των υδάτων. Το 12 πρόκειται προωθήθηκε μία ε, διάρθρωση με βάση το μπαμπού που επέτρεψε τη χορήγηση χιλιάδων ε, κυβικών μέτρων ύδατος. Το ίδιο ισχύει με τη, φωτοβολταϊκή και την αιωλική ενέργεια. Δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε σχέδια υπέρ του περιβάλλοντος που να ε, οδηγήσουν αυτές τις χώρες σε ανεξαρτησία σε σχέση με τους πόρους που διαθέτουν και θα μπορέσουν να διαθέσουν. Συνάδελφε, θέλετε, πολύ σωστά το θέμα των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Και είναι ένα μείζον πρόβλημα της ανθρωπότητας. Και έχουμε ευθύνη όλοι μας σε αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ευτυχώς η Ευρώπη είναι σε πολύ πιο ικανοποιητική θέση από τις άλλες περιοχές. Ξέρετε τα προβλήματα που έχουμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στα θέματα εκπομπών, αερίων και όλα αυτά. Και θα έλεγα ότι ως Ευρωπαίος νιώθω σε συναντήσεις με ανθρώπους από άλλες περιοχές και παράγοντες πολιτικούς πολύ πιο καλά διότι εμείς τουλάχιστον έχουμε μια πρωτοποριακή θέση σε αυτά τα θέματα. Και όντω οι κλιματικές αλλαγές είναι αυτές που φέρνουν τις φυσικές καταστροφές. Και στην Ευρώπη την ίδια. Οι μεγάλες κλίμερες που ζήσαμε στην κεντρική Ευρώπη. Αυτά που συνέβηκαν στα Βαλκάνια, στα Δυτικά τον τελευταίο Μάιο. Είναι αποτέλεσμα κλιματικών αλλαγών η υποσαχάρια Αφρική. Έχει όλα τα προβλήματα εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Που σημαίνει πρώτα ως Ευρώπη έχουμε μια ευθύνη να προωθήσουμε τις απόψεις μας σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με prevention, με πρόληψη. Αντιπλημμυρικά έργα στην Ευρώπη. Μέσω της βοήθειας ακόμη και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το σχεδιασμό που επιβάλλει στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προγράμματα που αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση, στη λογική του resilience building. Ότι στο Σαχέλ που έχει εναλλαγές πλημμυρών με ξηρασία θα πρέπει να οικοδομηθούν τρόποι να διαφυλάτεται υδάτινος σπόρτ για να αξιοποιηθεί την περίοδο της ξηρασίας. Όλα αυτά πρέπει να είναι στις μεγάλες μας στοχεύσεις πρέπει να είναι μέσα στα δικά μας πλάνα. Thank ευχαριστώ κυρία Χιμένες από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Κύριε Στυλιανίδη, θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί ε, θέτετε τα ε, θύματα στο επίκεντρο των μελημάτων σας για να τους ε, χορηγήσετε βοήθεια που χρειάζονται. Ως προς τα θύματα στην Ιγυρία ξέρουμε ότι η Μπόκο Χαράμ έδρασε αποτρόπαια απαγάγοντας αυτά τα ε, κορίτσια, κορίτσια για να δημιουργήσει ένα χαλιφάτο στη Βόρεια Νιγηρία. Υπήρξαν πολλοί εκτοπιστέντες, γι' αυτό θα πρέπει να χορηγήσουμε αρρωγή στα θύματα το ταχύτερο δυνατόν. Βεβαίως η φτώχεια είναι το αίτιο που οδηγεί στην ανάπτυξη της τομοκρατίας. Πώς θα αντιμετωπίσετε την πόκο Χαράμ λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολύ λίγοι διεθνείς παράγοντες που δρούν στην Ιγυρία γιατί υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Επίσης, ποια μέτρα θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε την την ανθρωπιστική πρόκληση όπου δύο εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες υποσυτισμού και υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στον κόσμο. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Έχετε δίκιο ότι η Νιγηρία παρόλο που είναι μια χώρα που θεωρείται σε επίπεδο ΑΕΠ ακαθάριση του εθνικού προϊόντος έχει το πιο σημαντικό πρόβλημα υποσυντισμού παιδιών. Δυστυχώ. Και η Πόκο Χαράμ, μια οργάνωση η οποία έφτασε όντω σε απαγωγέ κοριτσιών και έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Βόρεια Νιγηρία. Και δυστυχώ έχει 4.000 θύματα ήδη. Λοιπόν, αυτό που επιβάλλεται στην Νιγηρία είναι σε διαβούλευση με την ίδια την κυβέρνηση να πιστεί σε ό,τι αφορά τα θέματα του υποσυτισμού να περάσει στη διαδικασία του resilience building. Η Ευρώπη συνεισφέρει στα θέματα επισυντιστικής βοήθειας, αλλά μέσα στα πλαίσια της κατανομής του προϋπολογισμού θα πρέπει να πείσει την Νιγηριανή κυβέρνηση να γίνει πιο ενεργή στα θέματα του resilience building, της αθετικότητας. Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση και δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει εκτός της βοήθειας στην Ιγυρία και να συνεχίζει τη βοήθεια και στα παιδιά αλλά και στους πρόσφυγες εξαιτίας της δράσης της Μπόκο Από την άλλη, τα θέματα της πολιτικής λύσης, όπως είπα και πριν, είναι αυτά που θα δώσουν την τελική διέξοδο για να περιοριστούν τα ανθρωπιστικά προβλήματα. Αυτά είναι στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης και πώς θα δράσουμε ως project team με τον συντονιστικό ρόλο της κυρίας Μογκερίνη έτσι ώστε να βοηθηθεί η κατάσταση εντός της Νιγηρίας και σιγά σιγά να περιοριστεί ο ρόλος και η δράση της Μπόκο Γιατί είναι μια οργάνωση η οποία όντως φτάνει σε αυτά τα αποτρόπια εγκλήματα. Ευχαριστώ, επόμενος ο κύριος Σιλβα Περέρα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ στο δραματικό πρόβλημα των προσφύγων, γιατί βλέπουμε ολόκληρες κοινότητες που να χρειάζονται τη διεθνή αρρωγή άμεσα και αναπόδραστα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποδοτική αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και συνεργασία με όλους τους σημαντικούς εταίρους. Ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους είναι η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων ε, Εθνών για τους ε, πρόσφυγες υπό τον Αντώνιο Γκουτέρες που έχει προβεί σε μια αποφασιστική και αποδοτική δράση πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς στα διεθνή αυτά πλαίσια. Τώρα, ως προς τις ΜΚΟ και την εταιρική μας σχέση, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δεχτεί την συμπερίληψη των ΜΚΟ μέσα στα πλαίσια του προγραμματισμού της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και δράσης, που είναι ύψης της σημασίας για τις παρεμβάσεις που είναι απολύτως απαραίτητες. Θέτεται ένα μεγάλο ζήτημα που είναι και θέμα της επόμενης ανθρωπιστικής συνόδου στην Κωνσταντινούπολη. Η απόδοση και η αποτελεσματικότητα ανθρωπιστικής δράσης. Και πρέπει συνεχώς να αξιολογείται. Γιατί όντω υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι και είπα και πριν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και ο Επίτροπο και η Επιτροπή για να φτάσουμε σε κοινέ ευρωπαϊκέ θέσει για να μπορέσουμε μέσα στο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέχρι τη Σύνοδο να έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να πούμε. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Αντώνιο Κουτέρ, τον είπα το εκπρόσωπο για του πρόσφυγε, έχω ήδη μιλήσει μαζί του και έχουμε κουβεντιάσει διάφορα θέματα έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή αντίληψη. Ε, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην όλη διαδικασία και αντίληψη γύρω από το θέμα των προσφύγων. Πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλη η έκταση πλέον των προσφύγων από όλε τι ανθρωπιστικέ κρίσει που χρειάζεται ύψιστη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι πολύ καλή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι κοινώ παραδεκτό, αλλά έχουμε δυνατότητες ακόμη σε πρακτικά σημεία να, γίν, να βελτιωθούμε. Η κρίση στη Συρία και στο Ιράκ που τώρα είναι πολύ επίκαιρες είναι ένα σημείο που ο διεθνής οργανισμός, τα Ηνωμένα Έθνη και ο κύριος Γκουτέρες έχουν ένα ειδικό ρόλο και το συζητήσαμε αυτό στην περιοχή γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν το πιο κρίσιμο θέμα μέχρι την επόμενη συνάντηση. Το θέμα που έχει σχέση με, την, με τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη εντάσσεται και στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής αλλαγής που είναι ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί θα έχουμε ανάλογη συζήτηση. Thank you. Mr. Karski for the e Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρσκι από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και οι δύο οργανώσεις έχουν παρόμοιες απόψεις και σε πολλές περιπτώσεις και πολύ παρόμοια ατζέντα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κρίσεων, σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την διαμεσολάβηση και τις δράσεις μετά τις συγκρούσεις. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, όλα αυτά διοργανώνονται μέσω μια ειδική διαθεσμικής συμφωνία. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. πώ μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ και τι τμήματα τη διοικητικής αυτή και οικονομική συμφωνία μπορούν να επεκταθούν και να εναρμονιστούν. είναι όντω κοινώ παραδεκτό ότι είναι πολύ όντω σε ψηλό επίπεδο η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτηριστικά θα έλεγα το 40% της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάει σε οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το επίπεδο συνεργασίας υπάρχει και θεωρώ ότι ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό γιατί όντω υπάρχει μια εξειδίκευση, τεχνογνωσία και καλύπτει όλο τον κόσμο και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αποδεικνύεται ότι πρέπει αυτή η συνεργασία να κρατηθεί στο πιο ψηλό δυνατό επίπεδο. Και θα την κρατήσουμε και πρέπει να κρατηθεί. Το ότι χρειάζεται βελτίωση σε μερικά σημεία χρειάζεται. Το απέδειξε το πρόβλημα στην ΑΕΤ που αναφέρθηκε προηγουμένως. Εκεί υπήρξαν προβλήματα συντονισμού, υπήρξαν προβλήματα leadership, υπάρξει και ένα πρόβλημα accountability. Αυτά όντω θα πρέπει να συζητηθούν. Σα είπα και πριν, έγινε μια ήδη πρώτη επαφή με την πρόεδρο τη Ότσα, την κυρία Βάλερη Άμο, η οποία έχει αυτή την ευθύνη για την ατζέντα αυτή και πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση θα βρεθούν εκείνοι οι τρόποι αυτή η συνεργασία να, γίνει, να επικαιροποιηθεί, να γίνει ακόμα πιο επίκαιρη και να αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που αναφύονται εξαιτία τη έκρηξη τη ανθρωπιστική κρίση. Θεωρώ ω πάρα πολύ σημαντικό θέμα τη συνεργασία μα την ανέβρεση νέων χορηγών σε επίπεδο κυρίω χωρών του κόλπου και μουσουλμανικών κρατών που θα βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να δημιουργηθούν και οι κατάλληλε γέφυρες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε περιοχές που τώρα δεν υπάρχει. Thank you. Mr. Nart for the ALDE. Ευχαριστώ για την άλλη, κύριε Νάρσκ. Συγχαρητήρια κύριε ε, Στυλιανίδη γιατί ήσασταν πολύ ε, σαφής ε, και οι απαντήσεις σας ήταν ε, πολύ σημαντικές. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την έννοια της ε, κλεπτοκρατίας. Και η Γουινέα του Ισημερινού και η Νιγηρία υπόκεινται στο καθεστώς της ε, κλεπτοκρατίας, διότι πολλές κυβερνήσεις τι κάνουν, απορρίπτουν τις ευθύνες τους και τις αποδίδουν σε άλλους. Και θα ήθελα τώρα να μιλήσω για το Ισραήλ. Η Σύμβαση της Γενέβης ε, θεωρεί ότι αυτός που κατέχει ένα έδαφος θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες υγείας ε, και επιβίωσης. Δυστυχώς δεν το εξασφαλίζει αυτό το Ισραήλ. Και το Ισραήλ ε, βάζει τη λωρίδα της Γάζας σε έναν ε, εφιαλτικό κύκλο. Το 60% ε, των πόρων πηγαίνει στο Ισραήλ θα ζητήσουμε απόδοση ευθυνών από το Ισραήλ για τις καταστροφές έτσι ώστε να μην πληρώνουμε εμείς για αυτές τις καταστροφές και να πλουτίζουμε το Ισραήλ. Θα απαιτήσουμε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί διαφορετικά θα είμαστε και υποκριτές και ε, θα μας διέπει έλλειψη δραστηριότητας, πλήρης έλλειψη δραστηριότητας. σας λόγια και έχετε δίκιο ότι σε ό,τι αφορά κάποιες χώρες το πρόβλημα της διακυβέρνησης του Κάβερνας είναι ίσως από τα σημαντικότερα προβλήματα για να μπορέσει ακόμα και η ίδια ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, αλλά κυρίως να μπούμε σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια πρόκληση σε ό,τι αφορά την ολιστική μας προσέγγιση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε και αυτά στα πλαίσια του project team των εξωτερικών σχέσεων. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, νομίζω έχω δώσει τις σαφείς απαντήσεις. Ότι ναι, στην περιοχή Γάμα, όπου υπήρξαν τα σοβαρά προβλήματα κατεδάφισης υποδομών που χτίστηκαν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αίτημα της αποζημίωσης είναι δεδομένο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσβασης στη Γάζα. Μετά την εγκυχηρία φαίνεται ότι υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και έχουν πάει κάποιες αποστολές που αφορούν φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Η εγκυχηρία θα βοηθήσει να συνεχιστεί αυτή η πρόσβαση. η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων είναι ένα μέγα θέμα και ξέρουμε όλοι μας ότι η Παλαιστινιακή κρίση είναι μια κρίση που δημιουργεί παγκόσμιες ανακατατάξεις, παγκόσμια προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη θέση. Την είπα και πριν με βάση την απόφαση της 30 Αυγούστου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιδιώκει τα δύο κράτη, ελπίζω στο πεντάλεπτο να το αξιοποιήσω για απάντηση απαντήσει ερωτήσεων. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βέντα από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε Επίτροπε για το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη φυσικών καταστροφών. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις περίπλοκων, πολύ περίπλοκων κρίσεων. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί τότε και με τις τοπικές κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα της ε, παροχής των ε, ανθρωπιστικών πόρων σε θέματα ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις κρίσεων. Η ανθεκτικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, όποτε δεν καταφέρνουμε να παρέχουμε βοήθεια, τουλάχιστον θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι μειώνουμε τον κίνδυνο του να συμβεί το χειρότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά η εταιρική σχέση και συνεργασία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, πολύ σημαντικές διαστάσεις. Τι πρόκειται να κάνετε λοιπόν για να υποστηρίξετε τις δράσεις των τοπικών κοινωνιών. Η μείωση κινδύνου καταστροφών είναι βασική αρχή του κύκλου της πρόληψης, του prevention και πρέπει αυτή η φιλοσοφία να επεκταθεί. Πρέπει πάση θυσία να ξεκινούμε από τη μείωση κινδύνου καταστροφών. Γιατί όπως είπα και πριν, το ένα ευρώ που δίνεις στη μείωση κινδύνου καταστροφών, στην πρόληψη, αντιστοιχεί με 4 έως 7 ευρώ την ώρα που θα, θα τα χρειαστείς για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και έχετε δίκιο ότι αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί αξιοποιώντα του τοπικού παραγόντε. Η κάθε περίπτωση όμω είναι διαφορετική. Παραδείγματο χάρη, το Αζίρ στο Σαχέλ ήταν διαφορετικό από το Σέαρ στο κέρα τη Αφρική. Ήταν διαφορετικό ο ρόλο των τοπικών παραγόντων στι δύο διαφορετικέ περιοχέ. Στο Νότιο Σουδάν, εκεί η πολιτική κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και τραγική που υπάρχει αδυναμία ακόμα και άσκηση του resilience building, όπως και στο Κόγκο. Που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο εύκολο πολλές φορές να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τον τοπικό παράγοντα, διότι υπάρχει η στοιχειώδης αδυναμία της πρόσβασης. Σημαίνει ότι η κάθε περίπτωση έχει αυτές τις διαφορετικότητες που θα πρέπει να τις λαμβάνεις υπόψη στον τρόπο εφαρμογής της φιλοσοφίας του resilience και της μείωσης κινδύνων καταστροφών. Θεωρώ όμω ότι η φιλοσοφία αυτή απεδείχθη στην πράξη ότι είναι η καλύτερη και μάλιστα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη, τον Επίτροπο Ανάπτυξη και όλε τι υπηρεσίε έχουν οδηγήσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είπα και πριν, εάν καταφέρουμε και κρατήσουμε το 20% ή και το επεκτείνουμε σε αυτόν τον τομέα, θα είναι πολύ σημαντικό. Uh, thank από τους σοσιαλιστές. Κύριε υποψήφιοι επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δέσμευσή σας για μια πολιτική όπου η Ευρώπη είναι υπερήφανη. Εκεί μπορούμε να επιδείξουμε πατριωτισμό και όπως είπε και ο Λουί Μισελ θα πρέπει να γίνει βιώσιμη και ορατή ιδιαίτερα για τους νέους που ψάχνουν ένα όραμα για την Ευρώπη. Ένα ζήτημα που το θίξατε μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε μεγάλος χρηματοδότης, 40% δεν είμαστε οι μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι χρηματοδότες ε, τους οποίους θίξατε και μιλήσατε για την Τουρκία, Ινδία, Βραζιλία, τις χώρες του κόλπου. Η δράση δεν είναι ίδια με τη δική μας, αλλά νομίζω ότι από πλευράς αποδοτικότητας χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Ας δούμε την ανθρωπιστική βοήθεια σε 10 χρόνια. Θα προωθήσετε αυτή τη συνεργασία και σε ποια βάση με αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι όντως στην καρδιά του προβλήματος των νέων χορηγών. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις έχουν τόσο αυξηθεί που δεν αντέχουν οι προπολογισμοί. Χρειαζόμαστε νέους χορηγούς. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες γύρω από τις χορηγίες. Αυτό συζητάμε και τα, και τα θέματα του κατεπιστεύματος, trust, τα trust funds. Όλα αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά ιδιαίτερα οι χώρες που είπατε, Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, χώρες του κόλπου, θα πρέπει να ενταχθούν στη μεγάλη προσπάθεια των νέων χορηγών. Είναι η μόνη δυνατότητα η ανθρωπιστική βοήθεια να κρατήσει το επίπεδό της. Αλλιώς δεν ξέρω αν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη ο νέος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δράσης να συνομιλήσει, να κινητοποιήσει παγκοσμίω αυτό το θέμα για την αύξηση των χορηγών. Θεωρώ και το επαναλαμβάνω μεγάλο στίχημα το summit στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι πολύ καλό και συμβολικό το ότι γίνεται στην Τουρκία. Και θεωρώ ότι στέλνει μηνύματα πολλά πολιτικά που έχουν σχέση και με τις μουσουλμανικές χώρες. Και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Και στη διάρκεια της προετοιμασίας για το Σάμιτ, αλλά και στο ίδιο το summit. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Πώς θα αυξηθούν οι χορηγοί για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Θα πρέπει να βρεθούν και άλλες λύσεις. Είπα πριν για τα κατεπιστεύματα, τα trust funds. Θα πω και κάτι που έχει σχέση με τη συνεργασία χωρών, member states με την ΕΚΟ. Ήδη στην αχτή Ελεφαντοστού έχουμε μια άμεση χορηγία από πλευρά Γαλλία μέσω τη ΕΚΟ για να δοθούν λύσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξελίσσεται κάτι με τη Βρετανία, γύρω στα 140 εκατομμύρια. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. E ευχαριστώ κύριε Ζέλεφ από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε μου άρεσε πάρα πολύ η πρόταση που μας ε, γράψατε εδώ πέρα ότι δεσμεύομαι να βοηθήσω τις ξεχασμένες κρίσεις όπου ο λαός που πλήττεται και υποφέρει δεν προβάλλεται πλέον στη δημοσιότητα. Και είχατε πει ότι το πρώτο σας ταξίδι θα γίνει στις περιοχές ε, του έμπολα. Αυτό λοιπόν είναι στη δημοσιότητα, αλλά το Νότιο Σουδάν δυστυχώ που αναφέρατε δεν προβάλλεται στη δημοσιότητα. Πριν από τρία χρόνια ο κόσμο με, μεγάλη με ενθουσιασμό γιόρτασε την εξαρτησία τη χώρα και εδώ και ένα χρόνο είναι πραγματικά ανθρωπιστική τραγωδία που διεξάγεται και παρά τις δυσκολίες θα λάβετε μέτρα προκειμένου οι εκατοντάδες χιλιάδες που φεύγουν και απειλούνται από πείνα να λάβουν βοήθεια από εμάς. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσόρισε την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν και είπατε σε πολλές περιπτώσεις ότι είστε πολιτικός επιτροπός. Ποια πολιτικά μέτρα λοιπόν θα λάβετε προκειμένου να συνεχίσουμε τις δεσμεύσεις μας και να βοηθήσουμε το λαό εκεί. Έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις ξεχασμένες κρίσεις στο έλεος τους. Και ενδεχομένως το Νότιο Σουδάν, εάν δεν συνεχίσει να τη χάνει βοήθεια να καταλήξει σε μια ξεχασμένη κρίση. Όμως έχω ενημερωθεί ότι για φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 50 εκατομμύρια για τον Νότιο Σουδάν μέχρι τον Ιούνιο, ακόμα 30 εκατομμύρια μέσα στο καλοκαίρι και τώρα αναμένονται άλλα 30 εκατομμύρια μάλιστα από το ε, αποθεματικό επίκουσα ανάγκη. Το σύνολο δηλαδή τη βοήθεια θα φτάσει τα 110 εκατομμύρια. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα. Δεν αφήνει τον Νότιο Σουδάν. Τώρα, σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Όντω δεν είναι τα αναμενόμενα. Υπάρχει ενδεχόμενο λοιμού στην περιοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα υποσυτισμού. Υπάρχει πολύ μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα πρόσβαση. Οι δύο αντιμαχόμενε παρατάξει δυστυχώς δεν επιτρέπουν ακόμα και την αξιοποίηση του πετρελαίου που είναι πλούτου για τη χώρα να είναι αυτή που θα βοηθήσει τη χώρα να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί μαζί με την, με την Επιτροπή Ανάπτυξης το resilience building. Υπάρχουν πολλά προβλήματα για να ασκηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική και να μπορέσουμε όντως να, να μπει το Νότιο Σουδάν σε μια λογική βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα κράτο που είναι στα τελευταία σε ό,τι αφορά τα θέματα επίπεδου ζωή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο ανθρωπιστής Ιάπωνας. Δυστυχώ, δεν μπορούν να υπάρξουν ανθρωπιστικές λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα. Πρέπει να βρούμε πολιτικέ λύσει. Και εδώ είναι ο ρόλο να βοηθήσουμε τον Νότιο Σουδάν να βρει μια στοιχειώδη πολιτική λύση. Παράλληλα με την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια που θα πρέπει να συνεχίσει, να μην γίνει ξεχασμένη κρίση. Σα um, um, Σας ευχαριστώ και μεταξύ των τελευταίων ερωτήσεων. Κύριε Σιλενίδη, έξι ερωτήσεις μένουν μόνο. Ο κύριος Ντάνς λοιπόν είναι υποεμονός από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, υποψήφια επίτροπε, αναφερθήκατε ήδη στην ε, κλιματική αλλαγή. Ασφαλώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το 2012 32 ε, εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν ε, λόγω φυσικών καταστροφών, 98% των οποίων οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος. Και φυσικά δεν συνδέεται κάθε ανθρωπιστική κρίση με το περιβάλλον και δεν είναι κάθε ανθρωπιστική κρίση που συνδέεται με το περιβάλλον που φτάνει στις ειδήσει. Βλέπουμε λοιπόν ε, στην Ασία ε, πλημμύρες, αλλού ε, ξηρασίες και το κλίμα αλλάζει υπερβολικά γρήγορα και ο κόσμος δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί αποτελεσματικά. Δεδομένης λοιπόν της αλλαγή του κλίματος και δεδομένης της πιθανότητας πρόκλησης περαιτέρω κρίσεων και ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια στην Επιτροπή Κλίματος και Ενέργειας θα συνεργαστείτε προκειμένου να τεθεί ένας σαφής στόχος για να ε, μειωθούν αυτοί, αυτές οι συνέπειες και να αυξηθεί η αρρωγή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ σταθερή και στέρεη. Γι' αυτό και στη Νέα Επιτροπή υπάρχει επίτροπος ειδικό για θέματα κλιματικής αλλαγής. Αυτή η πολιτική, εάν δεν συνεχίσει στο δρόμο που είπαμε, ουσιαστικά θα αυτοαναιρεθεί. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο, γνωρίζοντας μάλιστα, τουλάχιστον από πλευράς φυσικών καταστροφών, ότι βασική αιτία πολλών φυσικών καταστροφών είναι η κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να οπισθοδρομήσει στο θέμα των πολιτικών στην κλιματική αλλαγή. Ίσα ίσα φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει και άλλε μεγάλε χώρε να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση. Οι οποίε δυστυχώ μέχρι τώρα δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση στο θέμα τα περιορισμού εκπομπών αερίων και όλα αυτά. Σημαίνει ότι εμεί είμαστε σταθεροί και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και θα έλεγα να νιώθουμε και περήφανοι τουλάχιστον ότι είμαστε ίσω οι πρωτοπόροι παγκοσμίω. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Το δίδυμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε τις φυσικές καταστροφές από αυτή την κλιματική αλλαγή. Εμείς έχουμε δύο εργαλεία. Το ένα είναι η ανθρωπιστική δράση, το άλλο είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Και τα δύο αυτά εργαλεία ασχολούνται ακριβώς με την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Πολλές φορές είναι πολυτομιακές. Περιπτώσεις IT, Φουκοσίμα, οι οποίες ήταν εξαιρετικά μεγάλες. Ακόμα και ο τελευταίος τυφώνας στις Φιλιππίνες ήταν πολύ δύσκολη. Εκεί όμως ήταν παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και βοήθησε και στην Φουκοσίμα και στις Φιλιππίνες και στην ΑΕΤ. Στην ΑΕΤ υπήρξαν προβλήματα συντονισμού. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη εκεί για να συνεχίσει τη βοήθεια διότι. Tisztelt biztos jelölt úr, örömmel hallottam az előző válaszában, hogy kiemelt. Αγαπητέ Επίτροπε, με χαρά άκουσα ότι δώσατε ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπηρίες. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα αυτό. Θα γνωρίζετε ίσως ότι Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μοναδική, η μοναδική οργάνωση που έχει επικυρώσει την συνθήκη για τα δικαιώματα των αναπήρων. Και υπάρχει λοιπόν ένα εδάφιο στο κείμενο αυτό όπου αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις εμπόλεμων σειράξεων ή σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με αναπηρία. Ερώτηση λοιπόν, στο μέλλον πώς προτίθεστε να παρακολουθήσετε τον τομέα αυτόν. Και δεν μιλάμε μόνο για άτομα με αναπηρίες, αλλά σε περιοχές που μαστίζονται από πολέμους, μιλάμε και για άτομα που επηρεάζονται από αναπηρίες, τραυματισμούς και αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας όπου δεν λαμβάνουν επαρκή βοήθεια όταν πλήττονται από τέτοια προβλήματα υγείας σε περίπτωση πολέμων κρίσεων. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή να είναι προτεραιότητα και νομίζω προσφέρει αυτή την δυνατότητα και ένα νέο action plan που έχει σχέση με την υλοποίηση του consensus στα επόμενα χρόνια το πώς θα αντιμετωπιστεί η ευπάθεια, πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα βοηθήσουμε τις ευάλωτες ομάδες και ειδικά όλες αυτές που αναφέρατε. Είπα και πριν ότι υπάρχουν κάποιες, κάποιοι δείχτες και κριτήρια τα οποία έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων στα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει ακόμη και χρηματοδότηση ειδικών ορθοπαιδικών κλινικών παραδείγματος χάρη σε άτομα που από τις πολεμικές συγκρούσεις έχουν υποστεί προβλήματα που έχουν σχέση με την κινητικότητα ή άλλα. Νομίζω αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν. Και έχετε απόλυτο δίκιο και δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ πρόθεση αυτά να μην συνεχίσουν. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε σε πιο πρακτικό επίπεδο και σε βάθος χρόνου το πώς αυτές οι δείχτες και τα κριτήρια που έχουμε στα θέματα χρηματοδότησης και αξιολόγησης προτάσεων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα εντάξουμε νέες ομάδες ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους, θα πρέπει να είμαστε σε επαφή, να συζητάμε για να βρούμε αυτές τις λύσεις. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες που θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγηση αυτών των νέων δικτών και κριτηρίων για να γίνουμε ακόμη πιο επαντολεσματικοί στο θέμα της αντιμετώπισης και της βοήθειας προς τις ευάλωτες ομάδες. Thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Ο κύριος, ο κύριος από την ομάδα των Σοσιαλιστών. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, χαίρομαι ειλικρινά γιατί η προηγούμενη μεγάλη και αξιόλογη προϊστορία σας, πολιτική προϊστορία, δίνει κάποιες ελπίδες ότι θα αντιμετωπιστούν και τα θέματα των ανθρωπιστικών κρίσεων. Για να είμαι όμως ειλικρινής δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας γιατί αυτές οι κρίσεις και αυξάνονται σε αριθμό και πολλαπλασιάζονται και ταυτόχρονα αλλάζουν διαρκώς πεδία. Ε, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα στοιχίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ενώ προξενούν ανυπολόγιστες υλικές και οικονομικές καταστροφές. Συγχρόνως και δεν το αναφέραμε εδώ συχνά υπάρχει απειλή των ανθρωπογενών καταστροφών όπως για παράδειγμα τα πυρηνικά ατυχήματα που μάλιστα έχουν διάσων συνοριακές επιπτώσεις. Μήπως λοιπόν δεν είναι επαρκής ο νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να εξαντλήσετε την αναμφισβήτητη ευφυΐα και φαντασία σας στην εισαγωγή νέων θεσμών και στις δυνατότητες συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Είστε και καθηγητής φυσικής και γνωρίζετε αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη έχει αποκτήσει ήδη μια πολύ σοβαρή εμπειρία σε αυτά τα θέματα διότι με αίτημα της Ιαπωνικής κυβέρνησης συμμετείχε στην Φουκοσίμα και βοήθησε πολύ και αναγνωρίζεται αυτό. Είναι πολλά τα διδάγματα από τη Φουκοσίμα για αυτές τις καταστροφές. Γνωρίζω από την προηγούμενη μου θητεία ως κοινοβουλευτικό στην Εθνική Βουλή της Κύπρου ότι υπήρχαν προγράμματα που είχαν σχέση με τις πυρηνικές καταστροφές. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το ακουμπήσουμε ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας θεωρώ ότι ε, είναι μια είναι μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και πρέπει να τύχει επεξεργασίας ένα σχέδιο αντιμετώπισης. Από ό,τι έχω μάθει στην ενημέρωση υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης σε διάφορα επίπεδα αυτών των πολυτομιακών επιπτώσεων και καταστροφών. Στο θέμα του πυρηνικού ατυχήματος επαναλαμβάνω ότι η Φουκοσίμα έχει δείξει πώ μπορεί να είναι οι λεγόμενε παράπλευρε απώλειε και η επέκταση του φαινομένου. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός με πολύ καλή δομή. Θα επαναλάβω ότι ένιωσα περήφανο όταν με πήγαν στο ERCC, το κέντρο που, πάνω στο οποίο βασίζεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, γιατί είδα ότι η Ευρώπη, ναι, έχει ένα κέντρο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχτεί σε περιόδου έκτακτη ανάγκη. Ανά την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Σα λέω ότι το θέμα των πυρηνικών καταστροφών θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο συστηματικά και έχετε απόλυτο δίκιο. Um, Ευχαριστώ κύριε Στήρ. Επίτροπε, κύριε Υποψήφιε Επιτροπέ, πλησιάζουμε προς το τέλος της ακρόασης και Ακούσαμε πολλά για το επίπεδο των δεσμεύσεων και το πάθος θα έλεγα με το οποίο στρέφεστε προς τη δουλειά αυτή και θεωρώ ότι χρησιμοποιείτε και ικανότητες από την επαγγελματική σας κατάρτιση ως γιατρός όπου όταν δώσετε απαντήσεις, ε, ερωτήσεις. Για πείτε μας όμως τι γίνεται με την ε, στρατηγική επικοινωνίας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είστε δεσμευμένος για παράδειγμα να μεταβείτε στη Δυτική Αφρική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δέσμευση αυτή. Είπατε ότι θα καλέσετε γιατρούς να μεταβούν εκεί. Αλλά και αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν φόβους. Είναι λοιπόν απαραίτητο, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει και η σωστή επικοινωνιακή στρατηγική. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ρωτώ λοιπόν, πώς θα χρησιμοποιήσετε, πώς θα αξιοποιήσετε την εμπειρία σας, πώς θα αξιοποιήσετε τα προσόντα, τα επαγγελματικά για την ε, επικοινωνιακή πολιτική, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχετε δίκιο ότι τα θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής και visibility της δουλειάς της ανθρωπιστικής δράσης θα πρέπει να είναι σε πρώτο επίπεδο. Έχω την πεποίθηση ότι η προκάτοχος μου, η κυρία Γεωργίευα, ήταν πολύ καλή σε αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον παρακολουθώντας διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης στην προηγούμενη πενταετία υπήρξε πολύ σημαντικό visibility. Και αυτό ήταν καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη είναι πάρα πολύ καλό διότι το 15% πάει στι ξεχασμένε κρίσει. Αποδεικνύει ότι για εμά του Ευρωπαίου είναι ηθικό να μην είναι αυτό σκοπό το visibility. Και το κάνουμε πράξη. Όμω ε, πιστεύω ότι πρέπει να στέλνετε το μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι στηρίζουν την ανθρωπιστική δράση μέσα από δημοσκοπήσεις κατά 90% με 2 ευρώ τη μέρα από ό,τι φαίνεται και είναι έτοιμοι να τη στηρίξουν παρόλο που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση και αυτό αποδεικνύει το ήθος και το επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών, ότι συμμεριζόμαστε στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες του ανθρωπισμού. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία για τους εθελοντές θα βοηθήσει και σε αυτό το τομέα. Θα έχουμε μια ομάδα ανθρώπων, νέων ανθρώπων ενδεχομένω, οι οποίοι θα είναι οι πρεσβευτές της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας και δράσης παγκοσμίω. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα προσδίδει και visibility και θα στέλνει το μήνυμα και, στο, και εκτός Ευρωπαϊκού Σύνορου και εντός ότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι ανθρωπιστικές πολιτικές και βρίσκουν πρόσβαση στα θύματα παγκοσμίω για να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του εθελοντισμού θα είναι πολύ βοηθητική και στα θέματα επικοινωνιακής στρατηγικής. Thank η Πατρίσα Τόια από τους σοσιαλιστές ε, θα επανέλθω στον ιό έμπολα. Η επιδημία ε, στην ουσία επεκτείνεται σε χώρες που δεν έχουν ένα σωστό σύστημα υγείας ή έχει ε, καταστραφεί και δρούν ο Ερυθρός Σταυρός, οι γιατροί χωρίς σύνορα και άλλες μήκυο αλλά ε, δρούν και κυβερνητικές οργανώσεις ε, που απαρτίζονται από γιατρούς που μεταβαίνουν εκεί εδώ και δεκαετίες ε, και πάνε από σπίτι σε σπίτι. Όμως έχει καταστραφεί και αυτός ο ιστός υγείας. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός με τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επίγουσας βοήθειας. Ε, χαίρομαι γιατί και η κυρία Γεωργίεβα ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και επειδή τώρα θα ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό νομίζω ότι θα, μπορέσατε, θα μπορέσετε να πάρετε τη σκητάλη αλλά να συνεργαστείτε και με την κυρία Γεωργίεβα η οποία θα είναι υπεύθυνη επί ζητημάτων προϋπολογισμού κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς για να πάρω ένα πολύ σημαντικό know-how που απέκτησε και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ πετυχεμένο. Και πιστεύω ακράδαντα ότι ναι, είναι, θα δώσει πολλά εφόδια εάν με τιμήσετε με την έγκρισή σας για να μπορέσω να μπω σε αυτό το στίβο των μεγάλων των προκλήσεων που έχει η ανθρωπιστική δράση, γιατί είναι πολύ μεγάλος. Στον έμπολα, Είπα και πριν ε, ότι αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι ταυτόχρονα με την παρουσία γιατρών, νοσηλευτών και χτίσιμο κινητών μονάδων νοσοκομείων, θα πρέπει σιγά σιγά να αποκαθίσταται και ο μηχανισμός, ο ιατρικός μηχανισμός, τα ιατρικά συστήματα στις τρεις χώρες, Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε. Και είναι κατεστραμμένος δυστυχώ. Και αν δεν χτιστεί αυτός ο, ο μηχανισμός, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα. Απλώς αντιμετωπίσαμε το σύμπτωμα, όπως λέμε στην ιατρική δεν αντιμετωπίσαμε την ασθένεια. Η ασθένεια οφείλει να αντιμετωπίσει όντω και τα μεγάλα προβλήματα στα κατεστραμμένα συστήματα υγεία των τριών χωρών που έχουν δεχτεί τα πιο σοβαρά πλήγματα. Είναι παράλληλε ενέργειε. Άμεση ενέργεια στους, με του γιατρού παρόντε, αύξηση του ιατρικού προσωπικού, αύξηση νοσηλευτικού προσωπικού, κινητέ μονάδε, φάρμακα, αλλά την ίδια στιγμή και αποκατάσταση μέσω του Resilience Speaking και με τη βοήθεια του Επιτρόπου Ανάπτυξη ώστε να ξαναχτιστούν τα συστήματα υγεία. Είναι παράλληλε ενέργειε που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Δεν υπάρχει αφιβολία. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Και τέλο, τελευταίο. Έχετε την τελευταία ερώτηση να κάνετε. Κύριε υποψήφιε επιτρόπε, σας καλωσορίζω. Καλωσορίζω και την δέσμευσή σας, το πάθος σας και την προθυμία σας να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω την προθυμία σας να συνεργαστείτε με τον υποτε, υποτε εκπρόσωπο ε, και Επίτροπο για την Ανάπτυξη, κύριε Ντέβε, Μίθα, όπου προκύψουν προβλήματα. Μία ερώτηση λοιπόν τώρα δεδομένου του ξεσπάσματος έμπολα που δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε, που δεν μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε γέρος ε, τα απαραίτητα μέσα και δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε και την κρίση. Τώρα, πώς μπορεί να δράσει η Ευρώπη για να αναπτύξει νέα, νέα μέσα, νέες ικανότητες, για να συνεργαστεί καλύτερα, να συντονίσει καλύτερα και να προωθήσει και την διαλειτουργικότητα μεταξύ ημών και των άλλων παγκόσμιων φορέων, όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Ι.Π.Α. γιατί αποστέλνουν και στρατιωτικές δυνάμεις για να περιορίσουν την κρίση και διαλειτουργικότητα λοιπόν και σε ό,τι αφορά μεταξύ, τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και υπολείπων φορέων. θέσατε το πρόβλημα στην ολότητά του. Ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα συντονισμό όλων μας. Ο ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστική Δράσης είναι όντως να είναι μέρος αυτού του συντονισμού. Να κινητοποιήσει, να διατηρήσει την εγρήγορση, να έρθει σε επαφή με όλους τους φορείς, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Και ήδη στέλνουν συγκεκριμένα στρατεύματα ακριβώς για να στήσουν κινητές μονάδες νοσοκομείων. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι βασικοί donors Σκανδιναβοί, όλοι τα member states της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γίνει ένας συντονισμός. Πιστεύω ότι έχει ένα ρόλο ειδικό ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Δράσης σε αυτόν τον συντονισμό. Και θα πρέπει να τον επιδιώξει, να τον αναλάβει. Γι' αυτό που όταν ρωτήθηκα αν θα πρέπει να πάω, ναι, πιστεύω ναι. ακριβώ αυτό ο ρόλο όταν είσαι επί του εδαφου καταξιώνεται πιο πολύ. Στον προσφέρει ο αλλο διότι είσαι εκεί και ξερει το πρόβλημα άμεσα. Γι' αυτό αυτός ο ρόλος ο συντονιστικο θα αποκτήσει αξία όταν έχεις συγκεκριμένο ρόλο επί του εδαφου Επιμένω ότι είναι μια πέραν από συμβολική και πολύ πρακτική ενέργεια για να μπορέσουμε να μπούμε στο σωστό συντονισμό και να δρούμε παράλληλα και στα θέματα του resilience δηλαδή να βοηθούμε στην αποκατάσταση των συστημάτων υγείας, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και τις άμεσες ανάγκες σε επίπεδο γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά ακόμα και μηχανισμού, όπως υπόθηκε πριν, παραδοσιακού. Γιατί υπάρχει ένας παραδοσιακός μηχανισμός ιατρικής περίληψης στις περιοχές αυτές. Χρειάζονται να υπάρχουν φάρμακα, αποχέτευση, πόσιμο νερό, όλα αυτά είναι υπόβαθρο για να χτιστεί η διαδικασία της θεραπείας για ασθένειες όπως η έμπολα. Όλα αυτά χρειάζονται εμπειρογνωμοσύνη και επιτόπου προσέγγιση. Γι' αυτό η επίσκεψη έχει και αυτή την αξία. Well, uh, ε, Επίτροπε, έτσι ολοκληρώνει το γύρο των ερωτήσεων. Μιλήσατε και μας δώσατε υπερπλήρες απαντήσεις. Αν επιθυμείτε, έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε οτιδήποτε δεν προλάβατε να απαντήσετε και να κάνετε τα καλλιτικά σας ε, σχόλια. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά έχετε μέχρι πέντε λεπτά, ε, αν το επιθυμείτε. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από τρεις ώρες, νομίζω είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο και ανθρώπινο. Θα κλείσω με δύο κουβέντες ανθρώπινες. Γιατί νομίζω αυτά που είπαμε ήταν όλα και ειλικρινή και ανταλλάξαμε καθαρές κουβέντες. Αυτή είναι, εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θα πρέπει να είναι η βάση της συνεργασίας μας. Να μιλούμε ανοιχτά, σαν μια οικογένεια. Διότι αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και εσείς και εγώ, είναι πολύ μεγάλες προκλήσεις. Είπε πριν ο καθηγητής, δεν θα ευχόταν να ήταν στη θέση μου. Αλλά αφού μπήκαμε στην πολιτική με το πάθος της πολιτικής για να προσφέρουμε, είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε να προσφέρουμε. Θα πω όμως κάτι που έχει σχέση με το Κοινοβούλιο γιατί νιώθω κοινοβουλευτικός ξεκίνησε μια διαδικασία με τις εκλογές του Μαΐου, η οποία καταξίωσε την όλη εκλογική διαδικασία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση και με τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό το hearing σήμερα ήταν μέρος αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Και παρόλη την κόπωση που σας είπα πριν, εν τούτης το χάρηκα γιατί ήταν ακριβώς μια δημοκρατική διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία που καταξιώνει την πολιτική και στέλνει το μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά όργανα, δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά ο ένας του άλλου. Δεν στέλνουμε μεταξύ μας απλώς φιλοφρονήσεις. Κάνουμε πολιτική συζήτηση. Έχουμε πολιτικό διάλογο. Έχουμε διαφωνίε. Είπα μια διαφωνία που είχα με έναν συνάδελφο. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσει. Και είναι αυτό νομίζω το βασικό επίτευγμα όλη τη διαδικασία που ξεκίνησε από τον Μάιο και θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό θέλει ο Ευρωπαίος πολίτη για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην Ευρώπη. Και έχουμε και οφείλουμε να του το δώσουμε. Τελειώνω με το να πω απλώς ότι πήρα πολλά σήμερα από τη συζήτηση. Έχω πολλά ακόμα να μάθω. Πάρα πολλά να μάθω. Είχα μια πολύ καλή ενημέρωση από τους ανθρώπους της Γενικής Διεύθυνσης. Τον κύριο Σόρεσεν και την ομάδα του. Τον ευχαριστώ πολύ. 15 μέρες δεν κοιμηθήκαμε. Αλλά μάθαμε κάποια πράγματα γενικά. Τώρα είναι η ώρα να μπούμε στα εξειδικευμένα, στα πιο λεπτομεριακά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν μου δώσετε την έγκρισή σας, μαζί θα πορευτούμε και να μάθουμε περισσότερα όλοι μας, αλλά κυρίως να κάνουμε πράξη τις απόψεις μας και το έργο μας και να κρατήσουμε την Ευρώπη ως το βασικό χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας για να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Ευρωπαίοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στυλιανίδη για την ε, τελική σας, για τα καταληκτικά σας σχόλια. Χρειάζεστε ε, ξεκούραση και την αξίζετε. Οι συντονιστές θα συνέλθουν εδώ και κλεισμένων των θύρων, γι' αυτό θα ήθελα οι μη ενδιαφερόμενοι να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Μετά από την αποτίμησή μας θα αποστείλουμε μία επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων θα κλείσει τη διαδικασία ακροάσεων. Σας ευχαριστώ όλους που προσήλθατε, ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, γιατί υπερβήκαμε το χρόνο, το χρόνο μας. Καλό σας βράδυ.